Okay, colleagues. My apologies for my lateness. Can I go on to the... Καλημέρα σας συνάδελφοι, συγγνώμη για την καθυστέρηση και την καθυστέρηση αφήξή μου. Θα θέλω να περάσουμε τώρα στις αποφάσεις των συντονιστών κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης. Τώρα σε ό,τι τους διορισμούς των εισηγητών, ε, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου του κανονισμού 216 ε, τις ναυτιλιακές υπηρεσίες ε, ναι θα όντως ε, θα διορίσουμε εισηγητή τώρα σχετικά με την πρόταση κανονισμού αναφορικά με την εφαρμογή του, ε, του ενιαίου ευρωπαϊκού εθέρα το έλεγχο θα ορίσει συντονιστή. Τώρα για την απόφαση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου αναφορικά με την εφαρμογή τη ε, διαλειτουργικότητα τη ε, ΑΕΚΟ. Το ΙΑΛΔΕ θα χορηγήσει τον ε, εισηγητή και η πρόταση κανονισμού που τροποποιεί τον κανονισμό 103, μάλλον 1365 για τις θαλάσσιες Μεταφορέ και ομάδα των πρασίνων θα χορηγήσει τον εισηγητή. για την πρόταση της ΕΚΟΛ συμφωνήθηκε πως η Επιτροπή θα ζητήσει την εφαρμογή του σημαίνει διαδικασία στο άρθρο 49 και η ΕΚΟ θα ε, συντάξει την έκθεση τώρα για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας αποφασίστηκε να μην αναλυφθεί δράση και πρόταση αναφορικά με την Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ευρώπη για οι νέες διατάξεις αναφορικά με την εφαρμογή των πολλαπλών κύκλων και για το πρωτόκολλο του Λουξεμβούργου σχετικά με το θέμα του κινητού εξοπλισμού και ούτε εδώ θα ανελειφθεί δράση. Τα πρώτα του κανονισμού, ειδικά με το άρθρο 290 τη συνθήκη, αναφορικά με τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μια σειρά από νομικέ πράξει για τι ε, διαδικασίε με έλεγχο. Ε, οι συγητέ σχετικά με θέματα επιτροπολογία θα αναλάβουν. Τώρα την παρακολούθηση σχετικά με την ε, εκπομπή διοξιδίου του άνθρωπου που θα τροποποιεί την οδηγία 525. Οι πράσινοι θα αναλάβουν την ε, σύσταση, την συγκρότηση έκθεσης. Τώρα, επίσης σε ό,τι φορά τις μη δράσεις που, θα, που δεν θα αναλυφθούν, Υπάρχει πρόταση της, ε, του Συμβουλίου για απόφαση που θα πρέπει να αληφθεί από τις αρμόδιες επιτροπές του ΟΗΕ αναφορικά με κάποιους κανονισμούς και εδώ αποφασίστηκε ότι δεν θα αναλυφθεί δράση αυτήν την απόφαση των συντονιστών. Για τις κατευθυντικές πράξεις η απόφαση ήταν να συσταθεί, συστήσουμε στην επόμενη νομοθεσία να ορίσουν οι εισηγητέ για να παρακολουθήσουν τι κατεξόδου πράξει και κατά τη διάρκεια τη ε, ε, συνεδρία της, της επόμενης επιτροπής ε, του τρανς θα εξεταστεί είναι οι εξελίξεις τώρα επίσης το χρονοδιάγραμμα της ε, τραν θα αποφασιστεί και το θέμα της επιτροπολογίας σχετικά με τις επιστολές 24-26 κλπ το ζήτημα του FTL και αυτό θα διαβαστεί στους, στα μέλη το συντομότερο δυνατόν μόλις το λάβουμε. Αυτή είναι η έκθεση που είχα να σας κάνω σχετικά με τις δικαιές των συντονιστών και τις αποφάσεις που λάβαμε για τους ηγητές. Υπάρχουν σχόλια. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Ευχαριστώ πολύ. Ας περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Σε ό,τι φορά τον κανονισμό για τις ε, εξελίξεις των ε, διευρωπαϊκών δικτύων, εισηγητής ο κ. Κουμουτσάκος ε, και ο κ. Σέρτζοκ και η ψηφορία θα γίνει ηλεκτρονικός. Θα κάνουμε τώρα μια επαλήθευση, επαλήθευση έλεγχο δηλαδή, για να δούμε κατά πόσο λειτουργεί το μηχάνημα και κατά πόσο το ΕΛΚ δεν έχει υπεράριθμους βουλευτές. Ψήφισατε άπαντες, πέρας ψηφοφορίας. Δεν υπερβήκαμε τα όρια, εντάξει, καλή αρχή κάναμε. Λοιπόν, τώρα περνάμε στις πραγματικές ψηφοφορίες. Κουμουτσάκο Σερτούκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. 34 υπέρ 7 κατά 2 αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Κύριε Ερτούκ και κύριε Κουμτσάκο. Επόμενη ψηφοφορία. Πρόταση κανονισμού για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων είναι απόφαση για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Θα θυμόσαστε την ιστορία. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Α, έπρεπε να είχα πει ότι είναι του κύριου Κουν. 35-5. Εγκρίνεται. Κυρία Σενελόβα τώρα. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 37 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 2 αποχές. Και η τρίτη ψηφοφορία είναι της κυρίας Άφησαρ. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 37 υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές. Συνεπώς, οι εισηγητές έχουν την εντολή για διαπραγμάτευση. Και τώρα ερχόμαστε στην έκθεση Ντομινίκ Ρικέ Πρόκειται για τον εξοπλισμό πλοίων. Οδηγία 96-98. Υπέρ της τροπολογίας 35. Κατά αποχές ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36 και 37 που είναι ίδιες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Νομίζω ότι έχουμε την ίδια πλειοψηφία. Ελέγξουμε όμως καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β. Αλλά πού είναι η συμβαστική Α. Δεν τη βλέπω, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, συμβαστική Β υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41. αν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική, α, 47 καταπίπτει. Λοιπόν, συμβαστική γάμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 Πάμε στο άρθρο 13.1 αν εγκριθεί έτσι. 53 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 54, 55 και 57 μαζί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 56 με προφορική τροπολογία. Έχει κανείς αντίρρηση στην προφορική τροπολογία. Σας υπενθυμίζω συνάδελφοι ότι σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς πρέπει τρεις να έχουν αντίρρηση και όχι ένας μόνο προκειμένου η ένσταση να έχει ισχύ. Υπέρ λοιπόν. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε για την 62 παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας τη προφορίας. Απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε, νομίζω ότι είναι η ίδια πλειοψηφία με πριν, αλλά σε ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίες. Εγκρίνεται. Πώς το κάνατε αυτό δεν ξέρω, λέει ο πρόεδρος. Ας μην το ψάξουμε. Εγκρίνεται. 64 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική σιγματά φεφ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 72 και 73 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 28 και 76 που είναι ίδιες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 29 είναι γλωσσικής φύσεως. 77-78 81 και 82, 83, όλες αυτές. Ε. Μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 79 του κύριου Περνιό. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, ας ελέγξουμε για την 80 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις φοφορίες. Απορρίφθηκε. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε και για την 30. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε για την 33. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Η 1 και 2 μαζί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 34 υπέρ, κατά, αποχές. Ας ελέγξουμε για τροπολογία 34 παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε της φοφορίας. απορριφθηκε Απορρίφθηκε 21-21. Τώρα ψηφίζουμε την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε της φοφορίας. 37 υπέρ, 3 κατά, 3 αποχές εγκρίνεται. Και τώρα το ψήφισμα, υπέρ, ε, μάλλον ψηφίστε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της φοβορίας. 36 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. Και τώρα για τις διαπραγματεύσεις με την Ίντερ. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 41 ψήφοι υπέρ, 2 αποχές και κανείς κατά. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Δικέ. Okay, colleagues, we Εντάξει, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης. για το προϋπολεσμό του 2014 και σχέδιο παρουσίασης ε, η κυρία Λίχτεμπεργκερ θα εκπροσωπήσει την κυρία Ντιουράντ. Θα μεταφέρω το μήνυμα της ε, Ισαβέλας, η οποία δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Απλώς θέλω να περάσω τις διάφορες παραγράφους και να σας πω λιγάκι για τις προτάσεις που έχει υποβάλει η Ισαβέλα. Στην παράγραφο 1 προσπαθούμε να πάρουμε την πρόταση η οποία προήλθε από τη συζήτηση της ΕΜΣΑ και να βασιστούμε στις προηγούμενες αποφάσεις του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη ρήπανση από πλατφόρμες εξόριξης και ατυχήματα στη θάλασσα αυτό το θέμα λοιπόν που θίγει και η Υπηρεσία Ασφάλεια στη Θάλασσα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεπερνάει τα διάφορα θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε ω επιμέρου επιτροπέ, αλλά θεωρούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Η παράγραφο 2 αναφέρεται στην έλλειψη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πλευρών χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων και το συνδέοντα στην Ευρώπη. Εδώ θα καταθέσουμε μια πιο λεπτομερή τροπολογία από τη βάση των τελευταίων εξελίξεων για τις δημοσιονομικές προοπτικές, γιατί τότε που διατυπώθηκε αυτό το κείμενο δεν ξέραμε ακριβώς ποια ήταν η κατάσταση. Στην παράγραφο 3 αυτή, αυτή την παίρνουμε από την έκθεση για τις καινοτόμες τεχνολογίες για μια βιώσιμη κινητικότητα και αναφέρει τις ε, συνέπειες για τον προϋπολογισμό έρευνας και ανάπτυξης. Βλέπουμε λοιπόν εδώ να υπάρχει έλλειψη συγκεκριμένων δράσεων, κάτι το οποίο πρέπει να διορθωθεί. Η παράγραφος 4 δίνει ένα πιο συγκεκριμένο <laughs> χαρακτήρα στην ε, ηλεκτρική κινητικότητα που περιλαμβάνει τα τραμ, τα τρόλεϊ λοιπά Και όχι μονάχα τις αλλαγές που μπορούν να έρθουν στην ηλεκτροκίνηση των ιδιωτικών αυτοκινήτων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερη ισορροπία σε όλα αυτά τα θέματα για να εξασφαλιστεί μια ευρεία πρόσβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα στις πόλεις. Η παράγραφος 5 αναφέρεται στις προπαρασκευαστικές δράσεις για τον βιώσιμο τουρισμό και είναι η βάση για πιο συγκεκριμένες διατυπώσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού. Όλα αυτά μπορούν να μπουν στο, στην πρωτοβουλία κόσμε για τον τουρισμό που μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και φυσικά εγώ έρχομαι από μια τουριστική χώρα, επομένω όλα αυτά τα πράγματα με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορείτε να περάσετε, να μου δώσετε τις ε, παρατήρηση και να δώσω τα σχόλια αυτά στην Ιζαμπέλο. Κύριος Ρικέ, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ισαβέλα για την εργασία της. Πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα βρισκόμαστε στην ε, απαρχή ενός νέου δημοσιονομικού πλαισίου που θα <clears throat> ακολουθήσει μια πορεία ε, δύσκολη γιατί εδώ πέρα ξέρουμε ότι θα μειωθούν τα κονδύλια σε πολλούς τομείς και αυτό θέτει ιδιαίτερα προβλήματα ιδίως για τον τομέα των μεταφορών πέραν της διευκόλυνσης Connecting Europe όλος ο άλλος προπολογισμό θα μειωθεί κατά 8% περίπου κάτι το οποίο θα αλλάξει σημαντικά το τοπίο. Όπως μας υπενθύμησε η εισηγήτρια έχουν τεθεί σε συζήτηση ορισμένα θέματα, αλλά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε από μια πιο στενή έποψη προπολογισμού. Θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία <clears throat> αυτού του τομέα για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Είναι ένα τμήμα του προπολογισμού που έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και δεν έχει πάντα ληφθεί υπόψη αυτός ο χαρακτήρας του. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να υπογραμμιστούν στην ε, γραμμοδότησή μας όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το τέταρτο πακέτο συνδεδομικών θεμάτων θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Εδώ μιλάω για τις υποδομές στα πλαίσια του Connecting Europe. Είναι ανεπαρκής η χρηματοδότηση γιατί αν δούμε το προηγούμενο πλαίσιο η αύξηση σε τρέχοντα ε, ευρώ ε, 5 δισεκατομμυρίων <clears throat> είναι μονάχα αυτό το ποσό το οποίο προβλέπεται. Επίσης θα πρέπει να υπογραμμίσουμε περισσότερο το ρόλο των αποκεντρωμένων φορέων γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναδιάθρωση του έργου τους των αποκεντρωμένων φορέων, ανάθεση νέων καθηκόντων και θα πρέπει και η Κομισιόν και το Συμβούλιο να μας εξηγήσουν καλύτερα πώς μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε την πολιτική μεταφορών, να ε, επιφορτήσουμε αυτούς τους φορείς με νέα καθήκοντα Τα θετικά στοιχεία φυσικά αναφέρονται από την έκθεση της κυρίας Ντυρό, αλλά όπως είδαμε και στο τέταρτο σιδηροδομικό πακέτο, έχουμε ένα τεχνικό κομμάτι των προτάσεων αυτών που δίνει πολλές αρμοδιότητες και ευθύνες στον αρμόδιο αποκεντρωμένο φορέα, ενώ συγχρόνως μειώνεται ο προϋπολογισμός του. Τέλος, να σταθώ στα ερευνητικά θέματα. Ξέρετε ότι οι μεταφορές έτυχαν μεγάλων περικοπών μέσα στα ερευνητικά προγράμματα. Έχουμε κρατήσει περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ για το σύνολο των ερευνητικών προγραμμάτων. <clears throat> Θα πρέπει να αγωνιστούμε και στα πλαίσια των ετήσιων προεπολεσμών, γιατί η εμπροστοφόρτιση έχει ανάγκη να τονιστεί για να υπάρξει μετατόπιση των μεταφορών στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα βάλουμε υπόψη μας στο προπολογισμό, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών, όπως αναφέρεται στο πακέτο για τις αεροπορικές μεταφορές και που θα αντιμετωπίσουμε ως νούπο. Και επίσης θέλω να υπογραμμίσω το σημαντικό έργο της Επιτροπής μας για τα θέματα μεταφορών με στόχο καλύτερη υπηρεσία προς τον πολίτη, καλύτερη απόδοση. Όλα αυτά φαίνεται να βρίσκονται σε μετοπική αντίθεση με τις μειώσεις των προϋπολογισμών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκάρδια Ζαουλιάλ. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να προσθέσω κάποια σχόλια σε αυτά που έκανε ο κύριος Ρικέ για την γνωμοδότηση αυτή μεταφορών. Όπως υπογραμμίστηκε είναι σαφές ότι μετά την πολιτική ψηφοφορία που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο για το δημοσιονομικό πλαίσιο που είναι βέβαια πολύ περιορισμένο και όχι μόνο περιορισμένο αλλά έχει και ελάχιστα περιθώρια ελιγμών προκειμένου να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την χρηματοδότηση κάποιων πολιτικών που πιστεύουμε η Επιτροπή μας ότι είναι προτεραιότητα έτσι λοιπόν η δουλειά μας για τον παραπολισμό του 2014 θα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και αυτό πρέπει να αναφέρεται στη γνωμοδότηση. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε και διάφορα θετικά πράγματα για τα επόμενα χρόνια, κυρίως για το 2014 και αυτό είναι η συμφωνία στην οποία καταλήξατε και η κυρία Γιάλα και ο κύριος Ρικέ για την σύνδεση με την Ευρώπη, Connecting Europe. Να δούμε όμως πώς θα επηρεαστεί ο προπολογισμό από αυτές τις αλλαγές, δηλαδή τι κριτήριο διαλειτουργικότητας θα αποτελέσει μέρος του πρώτου στόχου και μέρος της χρηματοδότησης της μιας ή της άλλης γραμμής. Αυτές είναι μικρές αλλαγές. Αλλά πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας. Όταν προτείνει το προπολογισμό η Επιτροπή, δεν γνωρίζει βέβαια τι θα γινόταν με το Connecting Europe. Αυτό λοιπόν πρέπει να το υπογραμμίσουμε και να ελέγξουμε μέσω τροπολογιών στον προπολογισμό ώστε να πάει καλά. Τώρα πέρα από τις προτεραιότητες που ανέφερε η εισηγήτρια, πρέπει να αναφέρουμε και τα εναλλακτικά καύσιμα και υποδομές. Και αυτό είναι το τομέα προτεραιότητας για την Επιτροπή μας, τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι για τα επόμενα χρόνια. Έρχομαι τώρα στον τουρισμό. Εννοείται ότι στηρίζουμε το να παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα των πολιτικών μας στον τουρισμό. Συγχρόνως όμως πρέπει να απαιτήσουμε να υπάρξει γραμμή στον προπολογισμό με πραγματικές πολιτικές υπέρ του τουρισμού. Γιατί είναι μέρος των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να αρκεστούμε μόνο σε κάποιες προπαρασκευαστικές δράσεις ή πιλωτικά προγράμματα. Γιατί στο κάτω-κάτω αυτά έχουν αποδείξει την αξία τους ότι προχωράνε καλά Οπότε, άπαξ και υπάρχει μια επιτυχία σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, αυτό πρέπει να καταλήξει σε μια πραγματική πολιτική. Το τελευταίο μου σχόλιο, με λεπτομέρεια, Γιατί, γιατί πιστεύω ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε την γνωμοδότηση μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας στη Θάλασσα. Χρηματοδότηση χρειάζεται όπως χρειάζονται και πολλές άλλες Τέτοιε υπηρεσίε. Δεν θα πρέπει να είναι στην πρώτη παράγραφο δηλαδή της γνωμοδότησης κατά τη γνώμη μου. Είναι θέμα, όχι βέβαια περιεχομένου, θέμα ε, μορφής, θέμα διατύπωσης. Να μην μπει στην πρώτη παράγραφο αυτό το σημείο. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Εγώ πιστεύω, μπορώ να διακριβώσω πόσο σημαντικά είναι τα προβλήματα που προέρχονται από τον προπολογισμό. Ξέρω ότι η Ιζαμπέλ δεν είναι παρούσα, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί της και πάλι. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια, ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ της όλο και μεγαλύτερης ευρωπαϊκοποίησης της πολιτικής μεταφορών με στόχο να υπάρξει μεγαλύτερη παροχή υπηρεσιών κινητικότητος, αλλά δεν έχουμε τα κονδύλια τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες κινητικότητας. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν περισσότερα χρήματα. Όλα αυτά έτυχαν υποσχέσεων, αλλά στην πράξη, μέσα στα πλαίσια των πολιετών δημοσιονομικών πολιτικών, προοπτικών υπήρξαν σημαντικές περικοπές. Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε, αν θέλουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, ότι θα υπάρχει η απόλυτη, η απαραίτητη χρηματοδότηση. Αυτό είναι το ένα σχόλιο μου. Δεύτερον, πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι το Συμβούλιο έχει κάνει ένα κατάλογο ονείων που είναι σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχει ζητήσει τη Παναγιά στα μάτια υπομορφή πρωτοβουλίων και αυτό δεν μπορεί να συνάδει με μια μείωση του προπολογισμού για του αποκεντρωμένου φορεί αναφέρθηκε ο φορέας για τα σιδηροδρομικά θέματα που έχει αυξανόμενη σημασία με το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο και έχουμε και την έμψα την υπηρεσία που έχει να κάνει με τη ρήπανση στη θάλασσα η οποία και αυτή πρέπει να έχει μεγαλύτερη αρμοδιότητα και για τις ε, πλατφόρμες εξόρυξης στη θάλασσα. Αυτό απαιτεί περισσότερο προσωπικό και όταν κάναμε τον έλεγχο των αποκεντρωμένων φορέων βλέπουμε ότι δεν βάζουν οποιονδήποτε σε αυτούς τους φορείς αλλά χρειάζονται ανθρώπους οι οποίοι να είναι πραγματικοί εμπειρογνώμονες και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ε, υποχρεώσεις τους και αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Για την καινοτομία και την έρευνα και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, ιδίω για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και την ε, βελτίωση των υποδομών για παραγωγή καθαρής ενέργειας Κάτι το οποίο εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η ηλεκτροκίνηση και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και στα πλοία να εξετάσουμε αντίστοιχες καθαρές μορφές ενέργειας και για τον τουρισμό φυσικά τη στιγμή που έχουμε μικρότερα χρηματικά ποσά είναι δύσκολο να επιτύχουμε τους στόχους μας είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε το βιώσιμο τουρισμό για τους πιο ηλικιωμένους και τα άτομα με ε, αναπηρίες και άλλα προβλήματα. Κατά τα άλλα νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Ο κύριος Μπράντμπερν. Ευχαριστώ. Πρώτον, όσον αφορά την γενική προσέγγιση της γνωμοδότησης αυτής. Ξέρετε, έχουμε δει τον τελευταίο καιρό ότι όταν έχουμε συνεδριάσεις του Συμβουλίου, αυτό που απασχολεί είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, οικονομική ανάπτυξη κλπ. Και πρέπει να πω, κοιτώντας τη γνωμοδότηση αυτή, δεν βλέπω τίποτα εδώ που να είναι στην πράξη ρεαλιστικό για να βοηθήσει τους στόχους αυτούς που επιθυμούν να πετύχουν όλα τα κράτη-μέλη και το διατυπώνουν στις διασκέψεις κορυφής. Η δεύτερη παράγραφος στη γνωμοδότηση αυτή είναι ένας κατάλογος ψευών πόθων. Το είπαν και οι συνάδελφοι από τους σοσιαλιστές. Οι προτεραιότητες εδώ δεν είναι οι προτεραιότητες που εγώ σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να έχουμε ως Επιτροπή Μεταφορών. Αν θέλουμε δηλαδή την οικονομική ανάπτυξη. Είναι πολύ ωραία να μιλάμε για ηλεκτρικά ποδήλατα κλπ. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι οικονομική ανάπτυξη. Άρα υποδομές που να λειτουργούν ικανοποιητικά και έτσι τα αγαθά, υπηρεσίες και οι άνθρωποι να μεταφέρονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πετύχουμε το στόχο της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς. Κάποια από τα θέματα τα οποία αναφέρονται εδώ μου φαίνονται περιφερειακά, Ποια σήμαντα. Είπανε και οι συνάδελφοι διάφορα για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι και τόσο ε, μεγάλος υποστηριχτής τους. Πάντως, πρώτη παράγραφος να λέει ότι θέλουμε τον προπολογισμό μας, ε, τουλάχιστον το σχετικό με τις μεταφορές, να πάει σε αυτήν την ε, υπηρεσία, δεν νομίζω. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί η γνωμοδότηση αυτή, να υποβάλουμε τροπολογίες έτσι ώστε οι μεταφορές να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη και δεδομένης της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αλλάξουν και οι προτεραιότητες. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόσμα τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Πού είσαστε. Α, εκεί ο κύριος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους και σας ευχαριστώ που κάνετε τη συζήτηση αυτή και στηρίζετε όπως συνηθίζετε την πρότασή μας. Θέμε σύντομος. Αυτό που θέλουμε να υπογραμμίσουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014 ε, ο προπολογισμό για τα μεγάλα προγράμματα μεταφορών θα είναι 6 φορές παραπάνω από το 2013. Ενώ λοιπόν βλέπουμε να γίνεται συζήτηση για τα σημεία που αναφέρατε κι εσείς, νομίζω ότι το σημείο κίνησης είναι πολύ θετικό δεδομένη της δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης. Για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς γνωρίζετε την πρόταση της Επιτροπής της 26 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τροποποίηση του προπολογισμού στις δημοσιονομικές αρχές για να αντιμετωπιστούν θέματα που έχουν να κάνουν με νέες αρμοδιότητες, με οργανισμούς κλπ. Ιδιαίτερα τώρα όσον αφορά την θάλασσα και τη ρήπανση, θα προτείνουμε για την ΕΜΣΑ ικανοποιητικό προπολογισμό τα επόμενα χρόνια για να αντιμετωπιστεί το θέμα της ρήπανσης των θαλασσών για τον ορίζοντα 2020. Εμείς, η Επιτροπή, πιστεύουμε ότι όλες οι πτυχές που αναφέρθηκαν εδώ και που είναι σημαντικές για την ανάπτυξη και την καινοτομία μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω του εργαλείου αυτού. Και από το 2014 και μετά θα μπουν στα βλάκια. Όσον αφορά τώρα την διαλειτουργικότητα και τα ευφύ συστήματα μεταφορών, έχουμε το Connecting Europe και έχουμε τη διευκόλυνση αυτή δηλαδή και έχουμε και τον ορίζοντα 2020 οπότε πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Με αυτές τις παρατηρήσεις σας ευχαριστώ που κάνετε τη συζήτηση και σας ευχαριστώ και για τη στήριξή σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ε, θέλετε να πείτε κάτι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα σχόλια. Θα τα μεταφέρω στην εισηγήτρια, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει η συζήτηση μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει κυρία Λιχτεμπέργια. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Η προθεσμία τροπολογιών είναι 24 Ιουλίου το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στις 5 Σεπτεμβρίου και Ολομέλεια δεν ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, 24 Ιουλίου είναι το μεσημέρι προθεσμία για τις τροπολογίες. Το επόμενο θέμα είναι το θέμα των ε, διπλωμάτων οδήγησης και η λειτουργικότητα των ε, ε, δυνατοτήτων. Η κυρία Τσικάου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εν συντομία, αυτή η οδηγία παρουσιάστηκε σαν πακέτο μαζί με τον κανονισμό που έχει να κάνει με τους ε, ψηφιακούς ταχογράφους. Και στις δύο περιπτώσεις ο στόχος ήταν να προωθήσουμε την ανάπτυξη των τεχνικών στοιχείων και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των ταχογράφων. Κατά την άποψή μου, η πρόταση της Κομισιόν ε, δεν λαμβάνει υπόψη όλες τις ε, πτυχές της ε, ε, ενσωμάτωσης των διπλωμάτων οδήγησης και της κάρτας οδηγού. Αυτό γιατί βασίζεται σε μια έκθεση αντικτύπου η οποία δεν λαμβάνει υπόψη αυτά τα στοιχεία και επομένως δεν είναι ικανοποιητική για μένα αυτή η πρόταση. Από την άλλη πλευρά ο κανονισμός για τον ψηφιακό ταχογράφο δεν περιλαμβάνει καμία ρήτρα που έχουν να κάνουν με την ε, ενσωμάτωση της κάρτας οδηγού και του διπλώματος οδήγησης. Το κοινοβουλίο μας ψήφισε σε πρώτη ανάγνωση για το θέμα του ψηφιακού ταχογράφου και ζήτησε να υπάρξει μια νομοθετική πρόταση αλλά με έκθεση σκοπιμότητας η οποία να αντανακλά όλα αυτά τα στοιχεία που έχει αξάρει το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να περάσει αυτό το πολιτικό μήνυμα ότι δηλαδή όταν η Κομισιόν παρουσιάζει τις μελλοντικέ νομοθετικές προτάσεις για τα θέματα αυτά, να ζητήσει το Κοινοβούλιο η έκθεση σκοπιμότητος να γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο και να λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές που έχουν να κάνουν με το εφικτό και τα ενδεχόμενα πλεονεκτήματα της συγχώνευσης της κάρτας οδηγού και του διπλώματος οδήγησης Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει μια ανάλυση όλων των τεχνικών δυνατοτήτων για μια λύση, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα συμβατικότητας των καρτών αυτών και η ασφάλεια των δεδομένων και η συμβατότητα των δεδομένων επιπλέον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ικανοποιηθεί από αυτή τη μελέτη αντικτύπου γιατί δεν έχει λάβει υπόψη το κόστος το οποίο θα προκύψει από αυτή τη συγχώνευση και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η, κατανο... η θέση από κοινού αυτών των, ψηφιακών πληροφοριών. Έχουμε τώρα σε πολλές χώρες τα Υπουργεία Εσωτερικών τα οποία δίδουν την άδεια ε, οδήγησης ενώ η κάρτα οδηγού δίδεται από το Υπουργείο Μεταφορών. Το να συνενωθούν τα πληροφορικά αυτά συστήματα και να χρησιμοποιούνται από κοινού, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνει η μελέτη σκοπιμότητος. Επίσης θα πρέπει να έχουμε κοινέ προδιαγραφές για, τις, ε, για τα ψηφιακά τσίπ των καρτών που θα πρέπει να υπόκειται σε κοινέ προδιαγραφές με τις άδειες οδήγησης. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να προβούμε σε μια εναρμόνιση όλων αυτών των προνοιών για τις κάρτες οδήγησης και τα διπλώματα οδήγησης. Η πρότασή μας λοιπόν είναι προς την Κομισιόν να ζητάμε μάλλον από τη δική μας Επιτροπή, την Επιτροπή Μεταφορών να απορρίψει την πρόταση της Κομισιόν και προτείνουμε να διενεργηθεί μια έρευνα, μια μελέτη η οποία θα παρουσιαστεί μέσα στα δύο επόμενα χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να υπάρξει τώρα χωρίς την κατάλληλη έκθεση αντικτύπου μια νομοθετική πρόταση αυτού του είδους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και αναμένω τα σχόλιά σας φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ την ε, επίοικιά σας Η κυρία Λίχτεμπέργκερ πρέπει να πάει στους, ε, στη Θεσμική Επιτροπή. Θα της δώσω το λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να πάω πράγματι στην Νομική Επιτροπή. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η κυρία Τικάου. Δεν είναι επαρκής η πρόταση της Κομισιόν. Δεν έχει την κατάλληλη έκθεση αντικτύπου. Η Κομισιόν προχωρεί πάντα προ τη δική τη κατεύθυνση ανεξάρτητα από τη θέση του Κοινοβουλίου και αυτό δεν είναι σωστό. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια διαθεσμική συνεργασία στα θέματα αυτά και νομίζω πραγματικά πρέπει να <clears throat> απορρίψουμε αυτή την πρόταση. ή να ασαφή σε πάρα πολλά θέματα, είτε πρόκειται για την προστασία δεδομένων, είτε την πολυπικιλία δεδομένων που βρίσκονται στα, στα τσίπ των καρτών στις ηλεκτρονικές αυτές κάρτες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι υπάρχει συνεκτικότητα της, στην πρότασή της δεν. Μπορούμε λοιπόν εμείς να ψηφίσουμε, να κάνουμε πρωτοβουλίες, να έχουμε πλειοψηφίες στο Κοινοβούλιο και στη συνέχεια η Κομισιόν δεν δίνει καμία σημασία στη θέση του Κοινοβουλίου. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα το οποίο έχει χαρακτήρα θεσμικό δεν μπορεί να υπάρχει μια πρόταση της Κομισιόν η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Η Κομισιόν λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την άποψη των άλλων θεσμικών οργάνων και εάν δεν το κάνει αυτό θα πρέπει να απορρίψουμε την πρόταση αυτή και να σου πούμε ξαναρχίστε και πάλι από την αρχή. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί υπάρχει μεγάλο ποσοστό απατών στον τομέα αυτό αν θέλουμε να έχουμε λοιπόν μια εμπεριστατωμένη πρόταση, τότε χρειαζόμαστε μια πραγματική έκθεση αντικτύπου. Εμείς είπαμε τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η έκθεση αντικτύπου, γι' αυτό πιστεύω ότι η καλύτερη αντιμετώπιση από τη δική μας πλευρά είναι η απόρριψη πρόταση της Κομισιόν. Και σας ευχαριστώ. Κύριος Κοχ. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να υποστηρίξω την κυρία Τικάου και να την ευχαριστήσω για τα σαφή σχόλιά της. Και δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά τα οποία είπε. Δεν πρόκειται για ένα νέο δίπλωμα οδήγησης ή μια αλλαγή της οδηγίας που υπάρχει τώρα για το δίπλωμα οδηγού. Πρόκειται για την πρόταση της Κομισιόν να ενσωματώσει την κάρτα οδηγού που είναι απαραίτητη για τον ψηφιακό ταχογράφο στο δίπλωμα οδήγησης. Αυτό πρέπει να γίνει μονάχα μετά από μία έκθεση αντικτύπου. Είναι πάρα πολύ διαφορετικέ διαδικασίε για την αφαίρεση των διπλωμάτων οδήγηση στα κράτη-μέλη. Αυτά είναι θέματα που υπόκεινται σε εθνικέ αρμοδιότητε. Είναι πολύ δύσκολο να ενοποιηθούν και να εναρμονιστούν όλα αυτά. Γι' αυτό εγώ θέλω να υποστηρίξω απόλυτα την πρόταση τη ηγήτρια. Ευχαριστώ, κυρία Μάισνερ, ε, για του φιλελεύθερου. Σα ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Σίλβια Τικάου. Ξέρουμε ήδη από τις διαπραγματεύσεις για τον ψηφιακό ταχογράφο ότι τίθενται μένα πολύ σημαντικά θέματα και γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει μια εξισορροπημένη αντιμετώπιση για να δούμε τι απαιτείται για την εφαρμογή του ψηφιακού ταχογράφου. Η Κομισιόν προτείνει να ενσωματώσει πολλά πράγματα. Φυσικά υπάρχει τεχνολογική ε, καινοτομία αλλά πρέπει να σκεφτούμε, μπορούμε να ενσωματώσουμε και να συγχωνεύσουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την εξοικονόμηση κόστου, γιατί ο στόχο μα θα πρέπει να είναι να μειώσουμε το κόστο. Η Κομισιόν λέει, ότι αυτό μπορεί να είναι ελκυστικό για το, τους οδηγούς να κάνουμε αυτή την συγχώνευση, αλλά δεν λέει τι σημαίνει αυτό για τα κράτη-μέλη, για το τι Θεσμού και τι φορεί πρέπει να φτιάξουν τα κράτη-μέλη για τον καλύτερο έλεγχο. Και αυτό κατά πιθανότητα θα οδηγήσει σε πρόσθετο κόστο για τα κράτη-μέλη. Επομένως δεν νομίζω ότι υπάρχει μια σωστή εξισορρόπηση όλων αυτών των θεμάτων και η Κομισιό δεν έχει σκεφτεί σωστά όλα αυτά τα οποία λέει. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σωστό να, επανα... να απορριφθεί αυτή η πρόταση και να επαναφερθεί στην Κομισιόν. Επίσης υπάρχει και το θέμα της προστασίας δεδομένων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πάντα τίθεται σε όλες τις καινοτόμες τεχνολογίες Όσο πιο πολλά απλοποιεί κανείς, όσο πιο πολλά στοιχεία συγκεντρώνει, τόσο πιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος για τα προσωπικά δεδομένα να παραποιηθούν ή να ε, τύχουν ε, υποκλοπής κτλ. Αυτά λοιπόν για την κυρία Τικάου και εγώ την υποστηρίζω εξωρωμότητας των φιλελευθέρων. Η κυρία Φώστερ. Μερικά σχόλια να πω ότι συμφωνώ με την εισηγήτρια. Το είχαμε θίξει και εμείς εδώ και καιρό και είναι σωστό αυτό που λένε οι συνάδελφοι, ότι είναι εθνική αρμοδιότητα. Είναι πολύ περίπλοκο, είναι διαφορετικά κυβερνητικά σώματα, αρχές που ασχολούνται με αυτό. Οπότε εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι θα αποφεύγαμε τις απάτες αν υιοθετούσαμε μια τέτοια πρακτική. Αν συγχωνευτούν όλες αυτές οι άδειες σε μία, τελικά αν για, κάτι κάποια παράβαση και σου πάρουν την ε, άδεια οδήγηση, ε, χάνει και όλα τα υπόλοιπα μαζί. Το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη είναι σαφή. Φυσικά η τεχνολογία προχωράει online. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι στο μέλλον θα κάνουμε κάτι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν στις χώρες μας και δεν ταξιδεύουν από τη μία στην άλλη. Οπότε εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον ο οποίος κυκλοφορεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να αναγνωρίζεται η άδειά του από τις αρχές που μπορεί να τον σταματήσουν. Ε, σύμφωνοι. Ας δούμε όμως και τι γίνεται με τα χρήματα που πληρώνουμε για όλες αυτές τις μελέτες σκοπιμότητας. Κοστίζουν πολύ ακριβά, δεν είναι φτηνές. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν. Υπάρχουν άλλα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν κατά προτεραιότητα, όχι αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Ζαρικέ. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ την κυρία Τικάου για την εκθεσή της. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μου θυμίζει το ελικόπτερο του Λεωνάρντο Νταβίτσι. Είναι δηλαδή ένα σχέδιο εξαιρετικό για την εποχή του, αλλά με τα μέσα που διαθέτουμε σήμερα δεν θα μπορέσει ποτέ να πετάξει είναι αδύνατον ε, δεδομένης της κατάστασης της χώρες μέλη να εφαρμόσουμε αυτή την ιδέα, η οποία είναι πολύ ελκυστική, αλλά όχι ρεαλιστική. Ε, το είπανε λίγο πολύ όλοι. Η πρόταση λοιπόν που μας κάνει η συγγήτρια είναι απόλυτα λογική. Πρέπει να απορρίψουμε την πρόταση της Επιτροπής, της Κομισιόν. Ο κύριος Έλιμπερκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πολλοί υποστηρίζουν την ε, θέση της εισηγήτριας. Το έχετε διαπιστώσει κι εσείς φαντάζομαι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Τικάου βέβαια. Στα πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας για τον ταχογράφο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε την απροθυμία των συνομοθετών να εγκρίνουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα νέο άρθρο 27 στον κανονισμό. Το άρθρο αυτό έθετε την αρχή της συγχώνησης, της γόνευσης της άδεια οδήγηση με την κάρτα του οδηγού μέσω μιας πρότασης οδηγίας που θα οδηγούσε σε καλύτερα αποτελέσματα στους ελέγχους και εξοικονόμηση χρημάτων. Όμως, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμμερίζεται την άποψη των συνομοθετών, επειδή θέλουμε να δείξουμε πνεύμα συμβιβαστικό, συμφωνούμε με την διαγραφή του άρθρου 27 τελικά. 19 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποσύρει την πρότασή της που τροποποιεί την οδηγία για τις άδειες οδήγησης που αφορούσε τη συγχώνευση με τις κάρτες οδηγού. Η πρωτοβουλία αυτή είχε προταθεί ως συμπληρωματικό μέτρο και ήταν ανεξάρτητη από την αποδοχή όχι του άρθρου 27. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι η διοικητική διαδικασία αποσύρεται και θα αποσυρθεί και από την επίσημη εφημερίδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια και πάλι. Είναι δηλαδή η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση, για να είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα καλά. Ναι, ναι, σωστά καταλάβατε. Η Επιτροπή έχει πάρει αυτή την απόφαση, ναι. Καλώ, εισηγήτρια. Θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ε, αναφέρω και στην έκθεσή μου, ζητάμε την απόρριψη της ε, πρότασης ε, της Κομισιόν και όπως είπε η κυρία Μάισνερ, θεωρούμε πως η πρόταση αυτή θα πρέπει να αναδιατυπωθεί και να αποτελέσει αντικείμενο νέων συζητήσεων και πριν από μια ενδεχόμενη νέα πρόταση της Κομισιόν ζητάμε την ε, πραγματοποίηση μιας μελέτης αντικτύπου σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει το Κοινοβούλιο. Πάντω η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Κοινοβούλιο μα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η μελλοντική νομοθετική πρόταση θα περιλαμβάνει μια μπρέτα αντικτύπου, η οποία θα είναι κατάλληλα ε, γραμμένη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, για τα σχόλιά τους και είμαι πεπισμένη ότι το Κοινοβούλιο θα στείλει ένα μήνυμα πολιτικής φύσης κατά τις ψηφοφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο της μελέτης αντικτύπου όπως τελικά το επιθυμούμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να ακολουθήσω τις ε, το όλο τελετουργικό. 18 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία, το μεσημέρι και οι ψηφοφορίε για τα τροπολογιών και η, η έκθεση θα ψηφιστεί στην συνεδρίασή μα του Σεπτεμβρίου. Η επόμενη έκθεση είναι το ζήτημα των ε, <clears throat> εκτελεστικών πράξεων και των ε, και ζητάω από τους συγκητές Κούν και Αλκαμπάι να λάβουν το λόγο και έχει το λόγο πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μαζί με τον κύριο Αλκαντράου έχουμε συντάξει μια γνωμοδότηση για το θέμα αυτό, η οποία είναι στα χέρια των περισσότερων μελών της Επιτροπής μας. Έχουν υποβληθεί διάφορες ε, τροπολογίες. Οι μισές είναι δικές μας, από μένα και τον κύριο Καντράουι. Υπήρξαν τρεις τροπολογίες από την κυρία Γιάλα Σέντερ, η οποία επικρίνει την Κομισιόν γιατί αρνείται να έχει τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες διατηρούν τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εδώ συμφωνώ απόλυτα έχουμε και την απαραίτητη δυνατότητα για τον έλεγχο αυτό. Η κυρία Μάιστον επίσης ζητά από, το, ε, από την Κομισιόν να υποστηρίξει την άσκηση του ελεκτικού έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πάλι και αυτή εκφράζει τη λύπη της για την έλλειψη επαρκών ανθρώπινων πόρων. Βρισκόμαστε λοιπόν σε συμφωνία με αυτούς τους ε, συντάκτες τροπολογιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε, στους τομείς αυτούς να υπάρχει φυσικά μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Κομισιόν σε τεχνικά ζητήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά δεν θα πρέπει να έχουν ουσιώδεις πολιτικές σημασίες αυτές οι μεταφερόμενες, σημασία αυτές οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες. Και επίσης είναι απαραίτητο να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να αυτοελέγχεται η Κομισιόν. Πρέπει πάντα να υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπίσει το Κοινοβούλιο τις πράξεις αυτές εκχώρησης. Και είναι απαραίτητο να έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε πλήρως την εφαρμογή αυτών των πράξεων από την Κομισιόν. Συμφωνούμε με την τροπολογία 1 και θα την ενσωματώσουμε στην έκθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ελκαντραουή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ε, συνεισηγητή, βέβαια, τον κύριο Κιν. Μπορέσαμε να συνεργαστούμε πολύ καλά. Και εγώ θα είμαι σύντομος. Έχουν υποβληθεί διάφορες τροπολογίες που πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Συμφωνούμε με τις διάφορες τροπολογίες, μια μικρή μόνο αλλαγή μπορεί να θέλουμε. Και ο κύριος Κιούν και εγώ υπογραμμίζουμε διάφορα ζητήματα. Λέμε ότι το κοινοβούλιο μας θα πρέπει να μπορεί να εμπλέκεται και να συνομιλεί με τους ειδικούς από τα κράτη-μέλη σε ένα αρκετά προκαταρτικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Έτσι ώστε οι εκτελεστικές πράξεις να είναι πιο αποτελεσματικές και να μπορούμε και εμείς να επηρεάσουμε τις προτάσεις ε, που γίνονται προτού να είναι πολύ αργά. Δεν χρειάζεται εδώ να σας πω πολύ περισσότερα. Τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε περισσότερο χρόνο να μπούμε σε βάθος. Ελπίζουμε να υπάρξει ομόφωνα η υποστήριξη της πρότασής μας. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ και εγώ και τους δύο εισηγητές, τον κύριο Κούν και τον κύριο Αλχαντράουι. Έχουμε ήδη μια συσσωρευμένη εμπειρία τριών ετών με την εφαρμογή της Συνδίκης Λισαβόνας που δίνει ίσες εξουσίες στο Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο. Και η εμπειρία μας ήταν ότι δεν λειτουργούν πάντα τα πράγματα με το σωστό τρόπο. Η Κομισιόν πρέπει να είναι ο θεματοφύλακας των συνδικών, να κάνει προτάσεις και να εξασφαλίζει και την τήρηση των συνδικών. Λογικό είναι να θέλει να έχει τόσο δυνατόν περισσότερες αρμοδιότητες, αλλά συγχρόνως το θέμα είναι αν θα πρέπει να έχει αρμοδιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν λοιπόν δώσουμε εκτελεστικές εξουσίες στην Κομισιόν που δεν μας επιτρέπουν εμάς να έχουμε κάποια εμπλοκή ή όχι. Το θέμα είναι λοιπόν αν προτιμούμε εκτελεστικές πράξεις ή κατεχώρηση πράξης σε αυτή την περίπτωση. Πολλά λοιπόν θέματα φαίνονται ότι είναι τεχνικού χαρακτήρα αλλά πολλές φορές έχουν πολιτικές συνέπειες οι οποίες είναι μεγάλη σημασία. Όταν πρόκειται παραγωγικά για θέματα ε, ασφάλειας ή παραγωγικά θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει ως εκπρόσωπος των πολιτών της Ευρώπης το Κοινοβούλιο να συμμετέχει πλήρως και γι' αυτό νομίζω ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις διατηρούνται τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί είμαστε εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης και είναι ακριβώς αυτό το οποίο προβλέπει η Συνδίκη της Λισαβόνας. Γι' αυτό έχω καταθέσει μια σειρά από τροπολογίες με στόχο να ενισχύσουμε τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου και τονίζω και πάλι ότι η Κομισιόν ως θεματοφύλακας θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει την απαραίτητη πληροφόρηση και τις απαραίτητες γνώσεις και να έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών. Νομίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ όλων να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνει η Συνδίκη της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά το δημοκρατικό έλεγχο. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. προτού δώσω τον κύριο Κράμερ Έχουμε μια ομάδα επισκεπτών στην αίθουσα που, έχει προσκαλέσει από την κάτω Σαξονία η κυρία Μάιστερ. Καλώς ήλθατε λοιπόν στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω ότι θα σας διαφωτίσει και θα σας φανεί ενδιαφέρουσα αυτή η συνεδρία. Ακόμα και αν όχι, σας καλωσορίζω. Ο Μάικελ Κράμερ. σας ευχαριστώ και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να μιλήσω τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ομάδα επισκεπτών από την Γερμανία. Μα είναι από την κάτω Σαξονία, Μάικελ, όχι από τη δική σου περιοχή. Α, το ξέρω, το ξέρω. Είναι η πρώην Ανατολική Γερμανία βέβαια, αν σας έχει διαφύγει αυτό. Πάντα με τις ε, κατεχώρηση πράξεις εμείς έχουμε προσπαθήσει η Κομισιόν να βλέπουμε από την πλευρά μάλλον της Κομισιόν μία πρόθεση να περιορίσει τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Αυτό δεν έχει νόημα να το συζητάμε κάθε φορά που εμπλέκεται μία κατεχώρηση πράξη. Αυτό το είδαμε και με τη διευκόλυνση Connecting Europe. Πάντα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και έχουμε προσπαθήσει να έχουμε ε, συμβαστικές λύσεις για τα θέματα αυτά. Έχουμε δύο τροπολογίες για αυτό το λόγο, την 9 και τη 13 που έχουμε υποβάλει και εκπροσωπώ την κυρία Λίχτεμπερκ η οποία έπρεπε να πάει να ψηφίσει και αφορούν τα θέματα των κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων. Εδώ πρέπει να περιορίσουμε μονάχα στις διοικητικού χαρακτήρα πράξεις και ό,τι έχει πολιτικό χαρακτήρα δεν μπορούμε να το αλωτριώσουμε από το Κοινοβούλιο και να το δώσουμε στην Κομισιόν. Βέβαια δεν είναι πάντα σαφή τα όρια, αλλά εμείς ζητούμε και από την Κομισιόν με την τροπολογία υπαριθμών 13 να είναι συγκεκριμένοι σε σχέση με τα διαθεσμικά κριτήρια που θα πρέπει να πριτανεύουν για το διαχωρισμό μεταξύ κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων. Όταν μια έκθεση έρχεται ενώπιόν μας, θα πρέπει να είναι σαφές πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εξουσιοδότηση και πότε οι εκτελεστικές πράξεις. Εμείς ως ε, Κοινοβούλιο και ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας και δεν θα πρέπει να τα εκχωρούμε χωρίς να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Μάικελ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος ε, θέλει να λάβει το λόγο. Κάποιος από τους δύο συνεισηγητές για τα θέματα επιτροπολογίας θέλει να πει κάτι ή όχι. Κοβέρνερ. Εν συντομία για τον κύριο Κράμερ και την κυρία Λίχτεμπεργκερ. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει τη δυνατότητα αυτή στην ε, παράγραφο 292 σε ορισμένες περιπτώσεις να, φέρουμε την να δώσουμε, να εκχωρήσουμε την νομοθετική αρμοδιότητα στην Κομισιόν. Τα πράγματα δεν είναι τόσο σαφή όσο ήθελε ο κύριος Κράμερ βέβαια. Αναφέρεται ότι δεν πρέπει να έχουν ουσιαστικές πολιτικές συνέπειες. Αλλά τι είναι σημαντικές πολιτικές συνέπειες. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να το καθορίσει κανείς εξ αρχής αν κάτι πρέπει να είναι κατεχώρηση ή όχι. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να κάνει καμία σαφή διάκριση. Καταρχήν συμφωνούμε σε όλα αυτά τα θέματα. Από πολιτική άποψη δεν θέλουμε να δώσουμε εξουσία στην Κομισιόν, Έχουμε πάντως στις κατεχώρηση πράξη δυνατότητα να ανακαλέσουμε αυτή την εξουσιοδότηση μέσα σε ένα διάστημα τριών ε, μηνών, εάν παρακολουθήσουμε σωστά την εκτέλεση από την Κομισιόν. Μπορούμε να ανακαλέσουμε λοιπόν την εκχώρηση, αλλά το πρόβλημα είναι όταν ζητάει ένα θεσμικό όργανο να ελέγξει τον εαυτό του, η Κομισιόν συγκεκριμένα. Αυτό δεν μπορεί, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, πιστεύω. Τότε πρέπει να κάνουμε κάτι. Κύριε Αλκαδράου. Ναι, πρόεδρε. Ένα πράγμα θέλω να υπογραμμίσω εγώ. Υπάρχει τροπολογία για άλλα σέντερ που μιλάει για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην δικιά της πρόταση είναι μια σωστή πρωτοβουλία λέει ότι πρέπει η Επιτροπή να έχει τα αντανακλαστικά αφόρμητα στις περισσότερες προτάσεις να προτείνει στην αρχή της ε, διαδικασίας διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να προχωράει πολύ προσεκτικά. Διστάζει ε, για τις διαπραγματεύσεις, ενώ θα έπρεπε να θεωρείται ότι πιο φυσικό το να αρχίζουν διαπραγματεύσεις μαζί μας έγκαιρα θα πρέπει να είναι ένα δημοκρατικό αντανακλειστικό και να είναι πολύ περισσότερο από ό,τι βλέπουμε να είναι σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Υπενθυμίζω, ναι, για τα δημοκρατικά αντανακλαστικά, το σημειώνω. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα εδώ στις 5 Σεπτεμβρίου και στην Επιτροπή Νομοθετικών Υποθέσεων στις 14 Οκτωβρίου. Στην Ολομέλεια θα δούμε. Επόμενο θέμα. Είναι το τέταρτο πακέτο σιδηροδρόμων, τεχνικό θέμα. Πρόκειται για τρεις, τρία σχέδια εκθέσεων, Bilbao, Κράμερ και Ζήλε. Θα αρχίσουμε με την διαλειτουργικότητα. Είναι η κυρία Μπαραντίκα Θα ακολουθήσω το ίδιο σύστημα. Πέντε λεπτά οι εισηγητές, τρία οι και δύο οι υπόλοιποι. Οπότε σας παρακαλώ οι εισηγητές πέντε λεπτά ο καθένας. Θα σας είμαι ευγνώμων αν τηρήσετε έτσι το χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Την προηγούμενη εβδομάδα κάποιο που ταξίδευε προ το Στρασβούργο δεν μπόρεσε να φτάσει έγκαιρα στο ραντεβού που είχαμε μαζί γιατί το τρένο του με το οποίο ερχόταν έπρεπε να παραμείνει στο Λουξεμβούργο. Το Βέλγιο δεν έχει καταφέρει να αναγνωρίσει τα συστήματα σιδηροδρόμων που διαθέτει στο Λουξεμβούργο. Είναι, δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση αυτή. Έχουμε διαπιστώσει ξανά και ξανά ότι υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός και έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει κανείς ένα τρένο και να φτάσει φτηνά και γρήγορα από τη Βαλένθια στο Όσλο για παράδειγμα. Πρόκειται για τεχνικά προβλήματα, υποδομόνο, τα οποία θα μπορούσαν να ξεπεραστούν. Αλλά υπάρχουν και διοικητικά όμως προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα παλιά μονοπόλια που έχουν τα τρένα. Ο κατακαιρματισμός λοιπόν των σειροδρόμων στην Ευρώπη περιορίζει τη διαλειτουργικότητα του σειροδρόμου και δεν μπορεί να συνδυαστεί με οδικές μεταφορές ή θαλάσσιες ή ενέργειες. Και έτσι περιορίζονται οι δυνατότητες των χρηστών αυξάνεται το κόστος και μειώνεται και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας και έτσι δεν μπορούμε να πετύχουμε και τις επενδύσεις που θα θέλαμε, άρα περιορίζονται πολλοί δυνατότητες των επενδυτών που θα μπορούσαν όμως να γίνουν στον τομέα αυτών. Επίσης, θα μπορούσαν οι σιδηρόδρομοι να βοηθήσουν πολύ και την περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επιπλέον, οι δρομικές μεταφορές σήμερα εξυπηρετούν πάνω από 8 δισεκατομμύρια διαδρομές και μεταφέρουν 10% των εμπορευμάτων, πράγμα που σημαίνει 13, δισεκατομμύρια ευρώ και έναν ανατζήρο 73 δισεκατομμύρια και 800.000 θέσει απασχόληση. Στη Λευκή Βίβλο, στην οδικό χάρτη όσον αφορά τι ενιαίες μεταφορές στην Ευρώπη, μιλάμε Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το 2050 οι σιδηρόδρομοι θα πρέπει να αναλάβουν τις μισές εμπορικές μεταφορές και μεταφορές επιβατών μέσα στην Ευρώπη. Και έτσι πέρα από το ότι θα μειωνόταν το κόστος των μεταφορών και θα βελτιωνόταν η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των πολιτών θα μπορούσαμε να μειώσουμε κατά 60% τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα το 2050 σε σχέση με το 1990. Τώρα που σας παρουσιάζω την έκθεση αυτή δεν θέλω βέβαια να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες τις οποίες θα συζητήσουμε τους επόμενους μήνες. Θέλω όμως να μοιραστώ μαζί σας τη διάγνωση που γίνεται για την κατάσταση και τις συνέπειες που έχει η διάγνωση αυτή στις δυνατότητες κινητικότητας του πληθυσμού και στην ανταγωνιστικότητα. Γι' αυτό και προτείνω να εντοπίσουμε μαζί τις ατυχικές εκείνες που θα μας βοηθούσαν να λύσουμε τα κύρια προβλήματα τα οποία εμποδίζουν την Ευρώπη να έχει έναν ενιαίο σειροδρομικό χώρο. Και προσθέτω ότι για να ετοιμάσω την έκθεση αυτή ήρθα σε επαφή με 30 διαφορετικές υπηρεσίες και αυτή τη βδομάδα θα κλείσω τον κύκλο αυτών επαφών με τους χρήστες όπου θα συναντηθώ με άτομα με αναπηρίες και θα συζητήσουμε μαζί τι τροπολογίε θα μπορούσαν να υποβληθούν στην έκθεση αυτή. Οι περισσότεροι λοιπόν από του χρήστε συμμερίζονται την άποψή μου για την κατάσταση. Προσπάθησα να καταλήξω σε κάποιε λύσει αφού συζήτησα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μου λένε μάλιστα ότι είναι εφικτές οι λύσεις αυτές που προτείνω και λογικές. Όλοι πιστεύουν ότι οι σιδόδρομοι έχουν τεράστιο δυναμικό για το μέλλον. Για να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα νέο συνδρομικό χώρο στην Ευρώπη πρέπει να απλοποιήσουμε τις 11.000 τεχνικούς κανόνες μάλλον που ισχύουν στις διάφορες χώρες ε, μέλη και που απαιτούν άδειε από 28 διαφορετικές κρατικές αρχές οι οποίες στη συνέχεια πρέπει να περάσουν από άλλες υπηρεσίε με διαφορετικέ δομέ μέσα κλπ. Οι κανόνε επίσης δεν είναι και διαφανεί. και πολλές φορές διαπιστώνουμε μεγάλη αυθαιρεσία στην εφαρμογή τους. Η πολυπλοκότητα αυτή επηρεάζει βέβαια και την τυποποίηση και το να μπει σε κυκλοφορία το υλικό. Σήμερα το 10% του κόστου σχεδιασμού και διάθεση στην αγορά ενός σειρμού αντιστοιχεί στο διοικητικό ε, κόστος. Και αν πρόκειται να κυκλοφορήσει μόνο σε τρεις χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό φτάνει στο 30%. Και όλα αυτά μέσα σε έναν οικονομικό χώρο που θέλουμε να είναι ενιαίος και μάλιστα μετά από τρία πακέτα για τους σιδηρόδρομους που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι οι οδηγίες οι οποίες στον τομέα της διαλειτουργικότητας για παράδειγμα έχουν εγκριθεί, η 96-48 για παράδειγμα που έχει να κάνει με τις υψηλές ταχύτητες που συμπληρώθηκε με την οδηγία 2001-16 που έχει να κάνει με το ε, συμβατικά ευρωπαϊκά τρένα, και η οδηγία που έχει να κάνει με την διαλειτουργικότητα του 2008-57 δεν έχουν μεταφερθεί στα κρατη σε όλα τα κράτη-μέλη όπως θα έπρεπε. Με την νέα πρόταση λοιπόν πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε ρεαλιστικοί και να μειώσουμε το 20% του χρόνου που χρειάζεται μια νέα επιχείρηση για να μπει στην αγορά. Και συγχρόνως μειώνουμε και το κόστος που επιβαρύνει τον κατασκευαστή. Τα 50 δισεκατομμύρια που θα απελευθερούν έτσι τα επόμενα πέντε χρόνια θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή συνδρομική βιομηχανία και τη θέση της στην παγκόσμια αγορά. Για να γίνει αυτό, η έκθεση πάνω στην οποία δουλεύουμε δίνει μία συνταγή και αυτή είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Θα θέλαμε να πρόκειται για έναν γκισέ κατά κάποιο τρόπο που θα εκδίδει το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο των ε, Τρένων. Πιστεύουμε ότι έτσι μπορούμε να έχουμε μια πιο απλή διακυβέρνηση και να ενισχύσουμε το ρόλο του όταν πρόκειται για την εποπτεία των εθνικών ρυθμίσεων για να αποφεύγονται αντιφάσεις. Τέλος, θέλουμε να επικεντρώσουμε σε μία μόνο διαδικασία όλες τις ε, κατακαιρματισμένες διαδικασίες που είχαμε μέχρι τώρα για τις άδειε που δίνονται και για ε, το σταθερό εξοπλισμό έτσι όπως προβλέπονται στην Οδηγία 2008 του 57. Μία εναλλακτική λύση θα ήταν να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μητρό των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων, το οποίο θα τροφοδοτείται από τα στοιχεία που έχουν οι εθνικές υπηρεσίες. Ο Πρόεδρος, ολοκληρώστε κυρία Μπιλμπάου. Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό. Είναι περίπλοκο το θέμα και προσπαθώ να σας πείσω να προχωρήσουμε. Κυρία Μπιλμπάου, λέει ο Πρόεδρος, σίγουρα. Οι διερμηνείς όμως τα έχουν εξαντληθεί γιατί προσπαθούν να σας προλάβουν, μιλάτε πολύ γρήγορα. Οπότε ολοκληρώστε παρακαλώ. Ναι, θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι πιστεύουμε με όλα αυτά ότι δεν ε, γίνεται εδώ επικάλυψη. Θέλουμε η έρευνα και η καινοτομία να προχωρήσουν, να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα SIF to Rail. Όλες αυτές είναι προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες που έχουμε εμείς οι Ευρωπαίοι για τους ευρωπαϊκούς σιδηρόδρομους οι οποίοι μπορούν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην κινητικότητα των ατόμων και των εμπορευμάτων αλλά να βοηθήσουν και τη βιωσιμότητα. Θα έπρεπε λοιπόν να δούμε όλα αυτά τα θετικά των ε, τρένων και τις πολιτικές αποφάσεις οι οποίες δυστυχώς εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα των σιδεροδρόμων, τις επενδύσεις και την καινοτομία. Γι' αυτό και θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για τη γενοδορία σας. Thank you. Ευχαριστώ. Ευτυχώς έχουμε κάποιο χρόνο. Αλλά αν τα λέγατε αυτά χθε το απόγευμα θα είχατε φάει το σφυρί στο κεφάλι για το ΕΛΚ. Ο κύριος Ντεγκράντες Πασκουάλ. Εντάξει, τέσσερα λεπτά. Μπορείτε να έχετε τέσσερα λεπτά. Είμαι πολύ ανοιχτός και κυμπάρης σήμερα γιατί πλησιάζουν οι γιορτές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι είναι εύκολο να συμφωνήσουμε με το πάθος, με τα λόγια και το διαγνωστικό της εισηγήτριας διάγνωση μάλλον. Ενώ λοιπόν αυτή της φιλοδοξία θα πρέπει να δείξουμε μια κάποια ευελιξία ανάμεσα στην φιλοδοξία αυτή και το ενδεχόμενο του να λειτουργήσει και να εφαρμοστεί στην πράξη. Πιστεύω ότι από τα λόγια της διαπιστώνουμε ότι είναι αναγκαίο να εγκριθεί ένα νέο, μια νέα δέσμη συνδρομική η οποία θα πετύχει μια καλύτερη εναρμόνιση και η ανταγωνιστικότητα του του, του σύνδεσμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά έχω κάποιε εμβολίε αναφορικά με το σύνολο των μέτρων που προτείνει η Κομισιόν. Τώρα, το τεχνικό ζήτημα που μα απασχολεί τώρα αποτελεί βασίζεται μάλλον στην ασφάλεια και τη λειτουργικότητα και όλα αυτά συνδέονται με την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Η πρόταση της Κομισιόν λοιπόν, όπως και αυτή της εισηγήτριας, είναι φιλόδοξη και συμφωνούμε με πολλά από τα σημεία ε, με τον οποίο η Κομισιόν συμφωνεί αναφορικά με την ε, επικουρικότητα. Τώρα, ό,τι αφορά τώρα την θέση της εισηγήτριας ε, για την πρόταση οδηγίας, συμφωνούμε την ανάγκη να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες για οικονομική στήριξη των καινοτόμων τεχνολογιών που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα, καθώς επίση του ορισμούς του άρθρου 2 και επίσης κρίνουμε ότι τη αμοιβαιότητα ανάμεσα στα κράτη-μέλη σχετικά με τις ε, τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Αλλά θα πρέπει να αξιολογήσουμε την ε, εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας στα άθρα 20 και 21 η πρόταση για την ε, θέση σε λειτουργία των ε, σειρμών αν πρόκειται για σειρμούς που λειτουργούν στο πλαίσιο μιας χώρας τότε θα πρέπει να υπάρχει αυτή η κοινοποίηση των εθνικών οργανισμών αλλά και των ευρωπαϊκών οργανισμών. Θα πρέπει τώρα το να έχει κανείς την μόνιμη, ε, μόνιμο έλεγχο και εποπτεία των διαφόρων υποδομών είναι κάπως επικίνδυνο. Θα πρέπει λοιπόν οι εθνικές αρχές ε, να εξοδοτούν την εφαρμογή των, σύστημα, των ελέγχου και σήμανσης, ε, σηματοδότηση μάλλον περίπτωση αυτή θα μπορούσε να υπάρξει μια ειδική ρύθμιση για τους εθνικούς ε, ρυθμιστές και αρχές. Τώρα, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ε, περαιτέρω φιλόδοξη, ε, ιδιαίτερα φιλόδοξη, θα πω ότι η συγκίδρια είναι περισσότερο. Είναι έτη περαιτέρω φιλόδοξη από την συγκίδρια σχετικά με τη θέση σε ισχύ αυτής της οδηγίας κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ένα μεγαλύτερο άχθος όχι για τις εθνικές αρχές αλλά και για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σύνδρομων. Αυξάνονται οι αρμοδιότητες και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο περισσότερο προσωπικό, καλύτερη κατάρτιση αυτού και κατά λίγο πρόεδρος, πρόεδρε μεταξύ το σύνολο λοιπόν των προτάσεων για το τέταρτο συνδρομικό πακέτο είναι πραγματικότητα και έκανε μεγάλες προσπάθειες η Κομισιόν αλλά και η Συγήτρια με την οποία θέλουμε να συνεργαστούμε για να αυξήσουμε την προσθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Μια μεγαλύτερη φιλελεύθερη του της δέσμης και που κατακλείδει η Πρόεδρε θα οδηγήσει σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με διαφάνεια και καλύτερη παροχή υπηρεσιών στον Ευρωπαίο πολίτη και Ευρωπαίους επιβάτες. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το ενδιαφέρον και την αφοσίωση που έχει δείξει για το θέμα αυτό. και πιστεύω ότι εδώ συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία με τρόπο ιδιαίτερα πεπλεγμένο. Και φυσικά υπάρχει το τεχνικό και το πολιτικό στοιχείο τα οποία συμπλέκονται. Και φυσικά η διαλειτουργικότητα είναι καταρχήν ένα θέμα το οποίο είναι τεχνικό αλλά και το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για να θέσει εμπόδια και σημεία αντίστασης από τους ιστορικούς φορείς μεταφορών στα κράτη-μέλη και από τις κυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν με το νέο αυτονομοθέτημα προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτή την αδράνεια και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε ώστε να υπάρξει μια εναρμόνιση ταχύτερη, να υπάρξει ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, να υπάρξει μια μεγαλύτερη λοιπόν δυνατότητα δράσης ώστε να ξεπεράσουμε αυτές τις ιστορικές αγκυλώσεις και αντιστάσεις, αλλά υπάρχουν και ορισμένοι ελοχεύοντες κίνδυνοι. Το γεγονός ότι ξεπερνάμε τους εθνικούς φορείς και προχωρούμε προς ένα ευρωπαϊκό φορέα, αυτό είναι πολύ σωστό, και το υποστηρίζουμε την ευρωπαϊκοποίηση της λήψης απόφασης στα θέματα αυτά, να υπάρξει ένα διαβατήριο με σε εισαγωγικά του τροχαίου υλικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά βλέπουμε ότι σε ορισμένε περιπτώσεις οι εθνικοί φορείς μπορούν να προτείνουν πιο σύντομο χρονοδιαγράμματα και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξισορροπήσουμε τα πράγματα, να καταλήξουμε σε μια κατάσταση καζάν-καζάν, δηλαδή να μπορούμε να έχουμε κέρδος όλων, θετικό άθροισμα. Να βοηθήσουμε τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Φορέα χωρίς να χάσουμε όμως την προσθέμενη αξία που μπορούν να μας δώσουν οι εθνικοί φορείς γιατί μπορούν να έχουν ταχύτερη επίτευξη αυτών των στόχων και με λιγότερο κόστος. Κάπου εκεί πρέπει να ψάξουμε λοιπόν να βρούμε την ισορροπία. Θα ήθελα τώρα να θέσω ένα ερώτημα προς την Κομισιόν ή προς τον αποκεντρωμένο φορέα για το αν θα μπορούσε να καταστεί δυνατό στη διαδικασία πιστοποίησης <clears throat> του τροχαίου υλικού και την εναρμόνιση αυτής της πιστοποίησης να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι οποίοι μπορούν να προχωρήσουν ε, ταχύτερο να είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τις γραμμές που έχουν το ευρωπαϊκό εύρος γιατί στην Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως ξέρετε υπάρχουν διαφορές από αυτό και επομένως εγώ πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να έχουμε και μια ομάδα εργασίας που θα δημιουργήσουμε για τη διαλειτουργικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία πρόσβασιμότητος στις υπηρεσίες όπως λέει και η συγγήτρια. Και τέλος θέλω να θέσω το ερώτημα μήπως για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την πρόοδο και να περιλάβουμε και τις απαραίτητες κοινωνικές πτυχές για τις οποίες αναφέρθηκαν και τα συνδικάτα για την πιστοποίηση του τροχαίου υλικού για συγκεκριμένους στόχους, αν μπορούν λοιπόν και οι κοινωνικοί εταίροι να παίξουν ένα μεγαλύτερο ρόλο και νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να τους χρησιμοποιήσουμε για μια βελτίωση της ποιότητας του τροχαίου υλικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τους πράσινους ο κύριος Κράμερ. Δεν μπορώ να σας τα πω στα ισπανικά και δεν ξέρω την κατάσταση στην Ισπανία αλλά έχουμε την κατάσταση που μετά από την Λισαβόνα μπορούμε να τα κάνουμε όλα με το αυτοκίνητο, με το αεροπλάνο, με το ποδήλατο κτλ. Αλλά με τα σιδηροδρομικά μέσα δεν μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Έχουμε πολλές διαφορετικές, πολλά διαφορετικά εύρη γραμμών στην Ευρώπη, τουλάχιστον 6 και 20 και παραπάνω διαφορετικά συστήματα σηματοδότησης. Πρέπει να υπάρξει μια απλοποίηση Φυσικά υπάρχει αυτή η τάση στην Ευρώπη και όλοι το βλέπουμε ότι είναι απαραίτητο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά υποκρύπτεται ο διάβολος μεταξύ των λεπτομεριών. Έχουμε τις εθνικές αρχές οι οποίες δεν κοιτάνε μακρύτερα από την εθνική τους μύτη και τα εθνικά τους σύνορα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τροποποιήσουμε. Τα συστήματα αυτά τα οποία έχουμε που είναι εθνικού χαρακτήρα οδηγούν σε καθυστέρηση και απώλεια χρημάτων. Αν θέλουμε εμεί να κάνουμε πιο εύκολη την κινητικότητα στην Ευρώπη και αν θέλουμε να προστατεύσουμε και το κλίμα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο ρόλο στις συνδεδομικές μεταφορές. Ξέρουμε ότι ένα, μια, μια ε, μηχανή σιδηροδρόμου η οποία είναι επιστοποιημένη σε μια χώρα μπορεί να χρειαστεί δύο ή τρία χρόνια για να αποκομίσει την απαραίτητη πιστοποίηση σε μια άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Και έχουμε πολλές φορές και το κόστος το πρόσθετο το οποίο προκύπτει. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μια μηχανή η οποία εγκρίνεται σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να εγκρίνεται να έχει αυτόματη έγκριση σε όλα τα άλλα κράτη γιατί αλλιώς το κάθε κράτος μπορεί να πει «Μα εγώ δεν το δέχομαι αυτό το όχημα γιατί έχει το α και το β πρόβλημα». Θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα συνολικό τρόπο πιστοποίησης. Προφανώς θα πρέπει να υπάρξει λειτουργία κοινή και συνεργασία μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών πιστοποίησης. Εμείς θέλουμε όμως και συμφωνούν όλοι οι εισηγητές ότι θέλουμε ένα κεντρικό φορέα, ο οποίος όμως θα συνεργάζεται με τους εθνικούς φορείς. Δεν θέλουμε ένα τεράστιο υδροκεφαλικό φορέα ο οποίος αντιμετωπίζει όλες τις λεπτομέρειες. Το μεγαλύτερο μέρος των ε, αποφάσεων θα πρέπει να λαμβάνεται ούτως ή άλλως από τις εθνικές αρχές. Αλλά πρέπει να υπάρχει ως πρώτος συνομιλητής ο Ευρωπαϊκός Φορέα Σιδηροδρόμων και αυτός θα πρέπει να συνεργάζεται με τι εθνικές αρχές. Αυτό δεν είναι καινούριο, το ίδιο πράγμα γίνεται και στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών υπάρχει ο Ευρωπαϊκός φορέα, ο οποίος έχει κάνει συγκεκριμένες συμφωνίες με του εθνικούς φορείς και σε περίπτωση ε, διαμάχης μπορεί πάντα να παρέμβει ο Ευρωπαϊκός Φορέας. Σε είναι η κατεύθυνση προς την οποία θέλουμε να κινηθούμε. Δεν θέλουμε να ε, πάρα πολύ μεγάλου μεγέθους ευρωπαϊκό φορέα ο οποίος θα αντικαταστήσει τις εθνικές αρχές. Για τις αρμοδιότητες του διαχειριστή υποδομών στην, ε, στα σιδηροδρομικά θέματα θέλουμε και οι βιομηχανικοί φορείς να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβουν και ένα μέρος της ευθύνης. Κανονικά δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Ένα αυτοκίνητο το οποίο παράγεται στην Ευρώπη μπορεί να κυκλοφορεί σε οποιαδήποτε ε, χώρα της Ευρώπης. Αυτό το αντίστοιχο θα πρέπει να γίνει και στα θέματα τα συνδρομικά. Να υπάρξει λοιπόν και η ευθύνη από την πλευρά των κατασκευαστών, αλλά και η δυνατότητα μιας ευρύτερης πιστοποίησης. Ο κύριος για τους ε, συντηρητικούς. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προετοιμασία, την εισηγητρία για το έγγραφό της και έχει φυσικά τονίσει τα θέματα τα οποία της είναι προσφυλή στην ίδια. Εγώ δεν θέλω να σταθώ τώρα στις λεπτομέρειες γιατί είχα την τιμή να συζητήσω, να παρουσιάσω, να συζητήσω στα πλαίσια της έκθεσης Κράμερ και να παρουσιάσω και τη δική μου έκθεση και επομένω δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που είπα. Το θέμα της διαλειτουργικότητος βρίσκεται πια σε στάδιο Οριμότητα, σε στάδιο πολιτικής συμφωνίας. Είναι σχετικά καλή αυτή η επιλογή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με το Συμβούλιο στα τεχνικά θέματα και εδώ θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένες πτυχές. Το ενίο σύστημα ε, καταγραφής και ταξινόμησης για τα οχήματα έλξης και για, τα, για το τροχαίο υλικό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν εμπόδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γιατί υπάρχουν αυτά τα εμπόδια. Θέλαμε να ξέρουμε ποιες είναι οι πληροφορίες από τον Ευρωπαϊκό Φόρεα Σιδηροδρόμων και πήγαμε και τους επισκεφθήκαμε για να τους ρωτήσουμε είναι σαφές ότι όταν πρόκειται για απομονωμένες αγορές σιδηροδρομικών υπηρεσιών δεν ξέρουν τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο να έχουν αυτές τις πληροφορίες. Υπάρχουν ε, γραμμές που είναι 1 και 52 και για αυτές τις γραμμές δεν έχουν αρκετές πληροφορίες στον Ευρωπαϊκό Φορέα σιδηροδρόμων. Αυτές οι πληροφορίες για να τις αποκτήσουν χρειάζονται να επομιστούν περαιτέρω κόστος για το πώς λειτουργούν. Επίσης για τις ε, μηχανές κίνησης υπάρχουν ε, μηχανές από τρίτες χώρες οι οποίες δεν διασχίζουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο συχνά και επομένως εδώ θα πρέπει να στοχεύσουμε στην μεγαλύτερη ευκαμψία και την πιο πραγματιστική δυνατότητα να έχουμε μια βάση δεδομένων που να καταγράφει όλες αυτές τις μηχανές σιδηροδρόμων. Δεν θα πρέπει να καταλήξουμε στο άλλο άκρο για τις απομονωμένες αυτές τις αγορές και να μειώσουμε τη δυνατότητα για τις ε, εταιρείε τρίτων χωρών να λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά όμως είναι λεπτομέρειες που μπορούμε να τις βελτιώσουμε. Εγώ δεν βλέπω προσωπικά να υπάρχουν μείζωνα εμπόδια τα οποία θα μας εμποδίσουν να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Περνάμε στα μέλη. Η κυρία Μέιζερ. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Μάσνερ. Η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων και των υπηρεσιών είναι κάτι το οποίο είναι ένας κοινό στόχος για όλους μας. Ξέρουμε ότι εγώ δεν συμφωνώ πάντα με τον Μάικελ, με τον Μίκαλ Κράμερ στα θέματα της ε, πολιτικής μεταφορών, αλλά συμφωνώ μαζί του όταν λέω ότι μπορεί να πάει κανείς παντού στην Ευρώπη με το πλοίο, με το άλογο, με το ποδήλατο, αλλά όχι με το τρένο. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια κοινή αγορά σιδηροδρομικών ε, υπηρεσιών και πρέπει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια τα οποία τίθενται σε επίπεδο ε, υπηρεσιών. Όταν βλέπω ότι έχουν δημιουργηθεί ορισμένες υποδομές ώστε να περιορίσουν την, ε, τον ανταγωνισμό, αυτό δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος. Είχαμε πολλά τέτοια προβλήματα στο παρελθόν. Έχουμε αυτά τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν οι εθνικοί φορείς για να εμποδίσουν την, ε, τον ε, ε, ανταγωνισμό. Όταν στη Βόρεια Ισπανία υπάρχουν τρία διαφορετικά εύρη γραμμών, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει άνοιγμα στον ανταγωνισμό. Εμείς λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Rail for Europe προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα των ε, γαλλικών και γερμανικών συνδρομών. Βλέπω τον κύριο Ρικέ ο οποίος υπομειδιά Μπορούμε λοιπόν με μεγαλύτερη συνεργασία να καταλήξουμε σε μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των εθνικών φορέων και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε ένα στόχο που όλοι μας υποστηρίζουμε σε πολιτικό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριο Σουπανιόν, έχει λόγο. Δύο λεπτά. Ζήλ, έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, το, θέμα της εξουδότησης ε, του τροχαίου λυκού είπαμε ότι είναι πολύ, ε, δημιουργεί πολλές καθυστερήσεις και αυτό επιδεινώνει την κατάσταση. Όπως είπε η εισηγητής, ε, συμφωνούμε με την ε, εισηγήτρια και θα πρέπει να υπάρχει νέος οργανισμός για την χορήγηση αδειών σύμφωνα επίση με την ανάλυση κομισιών σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης του συστημάτου αξιοδότηση και αδειοδότησης. Τώρα σε ό,τι φορά την αδιατύπωση αυτής της οδηγίας για τη διαφυλικότητα νομίζω ότι είναι ανεπαρκής. Ε, αντί να δούμε το σύνολο της κατανομής του νομοδιού ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία και την Υπηρεσία Ασφάλειας, θα έπρεπε να εξετάσουμε καλύτερα τις ανάγκες που προκύπτουν ε, για τις δυσκολίες που ε, έχουν δημιουργηθεί. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια ενιαία διαπαφή ανάμεσα στην Εθνική Αρχή Ασφάλειας και της εποπτείας της όλης λειτουργίας θα μπορούσε λοιπόν να οδηγηθούμε σε μια ενιαία αρχή για την αδειοδότηση και την, για τη δυνατότητα να ε, διέλθουν τουλάχιστον τα σύνορα μιας χώρας. Κατά τα υπόλοιπα, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ιδιωτόμων θα πρέπει να εμβαθύνει τα αποτελέσματα αυτή τη μεταρρύθμιση, όπω ανέφερε προηγούμενο, το θέμα τη ε, εκχώρηση ε, ε, δραστηριοτήτων και λειτουργιών στην υπηρεσία. διότι όλα αυτά θα πρέπει να ακολουθούνται από μια μεταβαρική περίοδο επαρκή που θα επιτρέπει μια ε, ρύθμιση των ε, νέων αυτών αρμοδιοτήτων. Γι' αυτό δεν μπορώ να υποστηρίξω πλοίο 66, 67 και 70, 69 και 70. Κύριος Γκρός. Πάρα πολύ σύντομα. Και εγώ θα ήθελα να δείξω αυτό το θέμα που ανέφερε η Γκεζίν Μάισνερ και ο Μικαελ Κράμερ δεν θέλω τώρα να μπω στις ε, ε, γενικές πτυχές των σιδηροδρόμων. Φυσικά υπάρχει μεγάλη δυνατότητα απασχόλησης από το βιομηχανικό τομέα και από την κατασκευαστική βιομηχανία στην Ευρώπη, η οποία απασχολεί περίπου 25.000 άτομα και το 1 τέταρτο των προϊόντων μας εξάγονται. Η Ευρώπη λοιπόν παίζει ένα παγκόσμιο ηγετικό ρόλο στα σιδηροδρομικά προϊόντα, αλλά περιμένουμε από την Κίνα και την Ιαπωνία να υπάρξει μεγάλος ανταγωνισμός. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα πρώτα απ' όλα να μπορέσουμε να δώσουμε τα απαραίτητα μέτρα και κονδύλια για την έρευνα, ώστε να μπορεί να υπάρξει μια ε, υποστήριξη της τεχνολογίας σε όλα τα κράτη και όχι μόνο η υποστήριξη τεχνολογικής ανάπτυξης μόνο σε ένα-δύο κράτη, Μα ενδιαφέρει από κοινού να κάνουμε τι βιομηχανίε και την έρευνα πιο αποτελεσματικέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια δεύτερη πολύ, πολύ σημαντική πτυχή είναι όχι μονάχα η έρευνα, αλλά η απασχόληση ατόμων που έχουν υψηλά προσόντα. Στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Πολωνία λείπουν οι τεχνικοί υψηλού επίπεδου. Αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι απαραίτητο αυτή η εκπαίδευση να βελτιωθεί, γιατί αλλιώ θα έχουμε πολλές δυσκολίες όταν αυτή η τεχνική θέλουν να πάνε από ένα κράτος στο άλλο. Επομένως αυτό σημαίνει μεγαλύτερη εναρμόνιση για την εκπαίδευση και την ε, αναγνώριση των δεξιοτήτων τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρώπη και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας όταν μιλάμε για τα θέματα αυτά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Θα δώσω το λόγο και στην Επιτροπή, αλλά προηγουμένως θέλω και εγώ να πω δύο λόγια. Αν σκεφτούμε σιδηρόδρομοι, έτσι, και ας ξεχάσουμε λίγο την πολιτική, παρόλο που είναι δύσκολο σε ένα κοινοβούλιο. Αλλά αν σκεφτούμε μόνο τους σιδηρόδρομους, οι τρεις αυτές εκθέσεις, που είναι τεχνικές, περιλαμβάνουν το πιο σημαντικό κομμάτι του πακέτου, γιατί αν δεν προσφέρουμε τη διαλειτουργικότητα, τα τεχνικά στοιχεία και την ασφάλεια, τότε τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε αυτά που λένε οι ευρωβουλευτές εδώ και για τις τρεις εκθέσεις. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό, πάντα μιλώντας σιδηρόδρομους μόνο, έτσι, γιατί εννοείται ότι μετά στις συζητήσεις με τις κυβερνήσεις και τα λοιπά μπαίνει και η πολιτική στη μέση. Αλλά αυτό που πρέπει να δούμε για αυτές τις τρεις εκθέσεις είναι πώς θα πετύχουμε την διαλειτουργικότητα. Όλοι το είπανε και ο Μάικλ και όλοι ότι Είμαστε στο 2013 και δεν είναι δυνατόν τα τρένα να περνούν τα σύνορα. Το 1969 ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι και το 2013 τα τρένα μας δεν μπορούν να περάσουν από μια χώρα στην άλλη. Εμείς στην Ευρώπη είμαστε στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την τεχνολογία των σιδηροδρόμων πρέπει να διατηρήσουμε τη θέση μας και να φροντίσουμε να έρουμε τους φραγμούς που υπάρχουν μεταξύ των χωρών μας, έτσι ώστε ως κλάδος να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλη την Ευρώπη. Τέλος, ξέρω ότι έχετε ακούσει αυτό που θα πω τώρα και άλλες φορές. Αν η πολιτική αεροπορία έχει τους ίδιους κανόνες που, έχει, που έχουν οι σιδηρόδρομοι σήμερα, τότε κανένα Airbus, κανένα Α380, κανένα 300 ε, κτλ. δεν θα πετούσε στην Ευρώπη. Θα έπρεπε να ζητούν πιστοποίηση, άδειε. Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε. Και πιστεύω ότι αν καταφέρουμε και ξεπεράσουμε τα τεχνικά ζητήματα και πετύχουμε τη διαλειτουργικότητα, έχουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, εννοείται χωρίς να κάνουμε καμία παραχώρηση στην ασφάλεια, εννοείται, τότε θα μπορέσουν και τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ να βρουν τη θέση τους. Αλλά αυτές οι τρεις εκθέσεις είναι ζωτικής σημασίας και για να επαναλάβω αυτά που είπε και ο Μάικλ, μην πάμε σε δύο χρόνια στο πέμπτο πακέτο και δεν ξέρω εγώ τι. Όχι. Εδώ είναι η καρδιά του ζητήματος κατά τη γνώμη μου, αυτές οι τρεις εκθέσεις. Λοιπόν, για πέντε λεπτά. Ο κύριος Πακέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που συμμερίζεστε τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το τόσο κρίσιμο κομμάτι του πακέτου. Ευχαριστώ την κυρία Μπιλμπάου για την παρουσίασή της και την έκθεσή της. οι συγγετές μερικές φορές είναι πιο φιλόδοξοι και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σωστά, πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Γι' αυτό και ευχαριστούμε για την έκθεση και τη φιλοδοξία της. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποια σχόλια επί των τροπολογιών. Πέρα από τη γενική αρχιτεκτονική που επιβεβαιώνει και την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία. Το ένα είναι εκεί που η συγγήτρια ενισχύει το ρόλο του οργανισμού όσον αφορά το EATMS. Το έχουμε ξανασυζητήσει και ξέρετε κι εσείς ότι η πτυχή αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες στο Συμβούλιο. Συμφωνώ πάντως με αυτά που ακούσαμε εδώ ότι ο οργανισμός θα πρέπει να αδειοδοτεί το ETMS ε αν θέλουμε να έχουμε πραγματικά διαλειτουργικότητα. Ευχαριστούμε λοιπόν για την τροπολογία αυτή, όπως επίσης και εκείνη που αναφέρεται σε ένα νέο μητρό καταχώρησης οχημάτων, προκειμένου να υπάρχει ομοιογενής διαχείριση των οχημάτων Ίσως πρέπει εδώ πέρα να σημειώσουμε και κάτι το οποίο δεν ακούστηκε πολύ σήμερα το πρωί, αλλά την προηγούμενη φορά ναι. Και αυτό είναι το θέμα των πόρων για τον οργανισμό. Θα υπάρχουν επιπτώσεις στους πόρους που δεν αναφέρονται ακόμα σε δήλωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά υποθέτω ότι όταν θα έχετε ολοκληρώσει εσείς το δικό σας έργο θα πρέπει να ξαναδούμε την δημοσιονομική δήλωση της Επιτροπής για ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της προσέγγισής σας. Το ότι συντομεύεται τη μεταβατική περίοδο, και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, πιστεύω ότι είναι πολύ καλό. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόσεξε πολύ και το ακούσαμε και στην ακρόαση ότι η μεταβατική περίοδος των τριών ετών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρκεί με το παραπάνω προκειμένου ο οργανισμός να εξοπλιστεί με ό,τι χρειάζεται για τις άδειες, γιατί στο κάτω-κάτω δεν μιλάμε εδώ πέρα για ένα μεγάλο Big Bang, μιλάμε για την αδειοδότηση. Θα μπορέσει λοιπόν να εκδίδει τις άδειες αυτές. Ένας χρόνος δεν είναι αδύνατον αλλά πρέπει να το δούμε βέβαια και στον διάλογο που θα αρχίσει με το Συμβούλιο για να δούμε τι θα πούνε και οι χώρες μέλη. Θέλω να σχολιάσω τώρα δύο πράγματα. Πρώτον, τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας για την διαλειτουργικότητα και την προσβασιμότητα που προτείνει η κυρία Γιάλα Σάντερ και το θέμα του ticketing για την προσβασιμότητα ο οργανισμός έχει ενημερώσει το STI. Αυτό τώρα θα εξεταστεί στην Επιτροπή RISK. Άρα θα υπάρχει ενημερωμένη νομοθεσία μέσα στη χρονιά. Θα καλύπτεται αυτό. Αλλά είμαστε στη διάθεσή σας κυρία Γιάλα να το συζητήσουμε αν θέλετε. Το ίδιο ισχύει και για το ticketing παρόλο που δεν έχει προχωρήσει αρκετά η δουλειά εκεί. Αλλά ευχαρίστω με τους συναδέρφους να τα συζητήσουμε αυτά παρατέρω. Για την επικορικότητα τώρα και τον ρόλο των εθνικών υπηρεσιών. Εννοείται ότι ο ευρωπαϊκός αυτός οργανισμός θα συνεργάζεται με τους εθνικούς, με τις εθνικές αρχές. Ίσως να υπάρξουν κάποιοι τομείς όπου οι εθνικές αρχές να παραμείνουν αρμόδιες, για τις υποδομές ίσως, όταν δεν έχει να κάνει με το ATMS στο Συμβούλιο μία προσέγγιση ήταν κάποιες αρμοδιότητες να παραμείνουν στις εθνικές αρχές. για το τροχαίο υλικό. Στα πλαίσια πάντως των ε, όσων αναφέρατε και εσείς και για να υπάρχει ένας ενιαίος δρομικός χώρος στην Ευρώπη, θα έχουμε λιγότερο εθνικό τροχαίο υλικό. Άρα οι ετούντες θα πρέπει πάντα να μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις εθνικές αρχές και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Τροχαίο Υλικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ε, οι συγητές, κύριε Μπιλβάου, θέλετε να επανέλθετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ε, ευχαριστήσω του συναδέλφου για τα σχόλια και θα αναφερθώ στα θετικά. Ναι, όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα βήμα για το ζήτημα της διαλειτουργικότητας και σήμερα στο, στον 21ο αιώνα όταν μιλάμε για καινοτομία, δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν ασχοληθούμε με, τρόπο, με θαραλέο τρόπο όλα αυτά τα ζητήματα θα παραμείνουν νεκρό γράμμα και θα χάνουμε χρόνο. Ευχαριστώ όλους όσοι είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουμε, είναι ένα καλό δείγμα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, το είχαμε ζητήσει και στην ε, έκθεση αρχικά, αλλά στη φάση της, ε, των τροπολογιών θα καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια για να μην, ορίσουμε, να μην ορίσουμε μόνο μία προθεσμία για τη μεταβατική περίοδο, αλλά έχουμε και ένα πρόγραμμα εργασιών, έτσι ώστε επειδή έχουμε ήδη μια εμπειρία με την ε, υπηρεσία αεροπορικών μεταφορών, να μπορέσουμε λοιπόν να συμφωνήσουμε όλοι. Ε, θα πω στον κύριο Ζήλε ότι και στον κύριο Γράμερ που είμαστε οι τρεις υπεύθυνοι για τις εκθέσεις, να δώσουμε λοιπόν μια συνοχή και συνέπεια στην όλη δέσμη και να εξάσουν θα γίνει με τις απομονωμένες περιοχές. Να πω στον κύριο Γκρός ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι ανταγωνιστική, αλλά θα πρέπει να αυξηθεί αυτή η ανταγωνιστικότητα. Έχουμε χάσει πολύ χρόνο με το ζήτημα των εξουσιοδοτήσεων των αδειοδοτήσεων και όλα αυτά κοστίζουν, διότι Υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις, χρειάζεται λοιπόν να βρούμε τη δυνατότητα να ε, υπολογίσουμε όλα αυτά τα ποσά, όλες αυτές τις δαπάνες για να πετύχουμε ένα θετικό βήμα. Χρειάζεται λοιπόν οι προθεσμίες να περιοριστούν, όπως είπα, να πω στην Κομισιόν ότι ε, Συμφωνώ με την αξιολόγησή τη. ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Αυτό το οποίο ζητάω είναι λίγο παραπάνω θάρρο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ο τομέα το χρειάζεται, υπάρχει ένα ζήτημα συναισθηματικό που αφορά στον φόβο. Θα ανοίξει η αγορά και όλοι φοβούνται τι θα, τι θα συμβεί με το τι με την ε, κατάσταση, διότι το άνοιγμα μπορεί να θεωρηθεί ότι θα πλήξει την εσωτερική αγορά κάθε κράτος μέλος. Αλλά πολλά θα χάσουμε αν δεν υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της Κίνας και της Ιαπωνίας που προχωρούν με ένα πολύ γρήγορο ρυθμό. Επίσης ε, είμαστε διατεθειμένοι διατεθειμένες καλύτερα διότι είμαστε μια ομάδα που αποτελείται από γυναίκες ε, και ευχαριστώ όλες και όλους για τις, ε, τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Ο κύριος Κράμερ είναι εισηγητής. 5-6 λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντική η ασφάλεια. Και αν συγκρίνουμε τι γίνεται σε επίπεδο ασφάλειας. Έχουμε 28.000 νεκρούς στην Ευρώπη από οδικά ατυχήματα, αλλά κάθε φορά που εκτροχιάζεται ένα τρένο γίνεται χαμός στα μέσα ενημέρωσης. Αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων στα, που μετακινούνται με σιδηρόδρομο ε, από 2 σε 3 εκατομμύρια το χρόνο, ενώ ο αριθμός των ε, θυμάτων από ατυχήματα κατέβηκε από 400 σε 100. Επομένως, είναι ε, απαραίτητο αν μιλάμε για ασφάλεια να μην οδηγούμε ποτέ αυτοκίνητο. Όλοι ε, αυτοί οι νεκροί βέβαια ακόμα και 100 είναι υπερβολικά πολύ, Αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι γίνονται μεγάλες πρόοδοι στα θέματα των, ε, της ασφάλειας και ζητούμε λοιπόν και από τους συνδεδομικούς φορείς και από τις αρχές ασφάλειας να κάνουν περαιτέρω βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Όταν λοιπόν υπάρξει ενοποίηση και εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Χρειαζόμαστε και στον χώρο της ασφάλειας να έχουμε ένα ευρωπαϊκό φορέα ο οποίος θα ελέγχει τα θέματα ασφάλειας και όχι να γίνονται αυτά μονάχα από εθνικές αρχές. Εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη συνεργασία μεταξύ των εισηγητών για τα θέματα αυτά, γιατί οι τρεις αυτές εκθέσεις, όπως είπε πολύ σωστά ο Μπράιαν, είναι εκθέσεις οι οποίες έχουν πολλά κοινά σημεία και πρέπει να προωθηθούν από κοινού. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε λοιπόν να υπάρχει μια ενιαία μορφή ελέγχου ασφαλείας και επιστοποίηση. και φυσικά όπως και είπα και στην προηγούμενη περίπτωση θα πρέπει να παραμείνουν οι εθνικές αρχές αλλά για την καλύτερη συνεργασία τους θα πρέπει να υπάρξει και ένας ευρωπαϊκός φορέας. Ο Μπράιν έθεσε το παράδειγμα των αεροπορικών συγκοινωνιών, το οποίο μπορούμε πραγματικά να μιμηθούμε και είναι πάρα πολύ σωστό. Όταν έχουμε λοιπόν μια ενιαία διαδικασία έγκρισης για τις ε, μηχανές έλξης, τότε αυτό θα οδηγήσει σε κέρδος για όλους γιατί θα είναι μικρότερο το κόστος, θα είναι μεγαλύτερη η δυνατότητά της να κυκλοφορήσει όλη την Ευρώπη. Και είναι σκανδαλώτης ότι δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα. Η... η ευθύνη βέβαια για όλα αυτά θα πρέπει να παραμείνει στους επιμέρους εθνικούς φορείς και θα πρέπει η εφαρμογή των εθνικών κανόνων να γίνονται με έναν τρόπο ο οποίος θα κοινοποιείται στον φορέα, τον ευρωπαϊκό. Έχουμε περίπου 12.000 συγκεκριμένες διατάξεις οι οποίες δεν εφαρμόζονται στην Ευρώπη, στον ευρωπαϊκό χώρο, εθνικές διατάξεις οι οποίες δεν εφαρμόζονται πάντα και αυτό πάλι είναι τρελό. Είναι απαραίτητο να υπάρχει η απαραίτητη κοινοποίηση από τις εθνικές αρχές και επανέρχομαι στην αρχή την, των, ε, της εποχής των σιδηροδρόμων ο ένας έβαζε φανάρια που ήταν μπλε και κίτρινα, ο άλλος κόκκινα και πράσινα και φυσικά δεν υπήρχε καμία λογική. Αν ήθελε κανείς να προειδοποιήσει παραδείγματος χάρη για μια φωτιά θα έπρεπε να είναι ενιαία όλα τα φανάρια τα οποία χρησιμοποιούνται για να δείξουν ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Είναι λοιπόν απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι η ασφάλεια δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως ένα οποιοδήποτε θέμα, αλλά είναι ένα ξεχωριστό. Για τις προθεσμίες μπορούμε πάντα να βραχύνουμε τις διαδικασίες πρέπει να ενθαρρύνουμε όλο το δυνατόν περισσότερο τις εθνικές αρχές να περάσουν σε ένα πιο σύντομο χρονικό διάστημα και βέβαια Υπάρχει πάντα η αντίρρηση από πολλού που λένε ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο προετοιμασία. Και επίσης θέλουμε να τονίσουμε και την ανάγκη μιας ε, κουλτούρας ασφάλειας. Όσοι έχουν ζήσει στο Βερολίνο ξέρουν ότι τα τραμ του S-Bahn στο Βερολίνο πάντα ουσιαστικά παραβιάσαν τους κανόνες εκεί. Αλλά εάν υπήρχε σωστή αστυνόμευση και εφαρμογή των κανόνων τότε η κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας ανώνυμος χώρος στον οποίο μπορεί ο κάθε πολίτης να λέει ναι εδώ υπήρξε παραβίαση των κανόνων και να μπορεί να διαμαρτυρηθεί χωρίς να υπάρξει καταδίωξή του στη συνέχεια. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε λοιπόν αυτές τις εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει στο παρελθόν. Έχουμε ε, φορείς, έχουμε ε, ατμομηχανές και μηχανές έλξης που χρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις αλλά δεν υπάρχει πολλές φορές ενίος ελεγχός τους. Επομένως, θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη χρησιμοποίηση των σιδηροδρόμων που είναι όπως είπα ένα πάρα πολύ ασφαλές μέσο συγκοινωνίας να χρησιμοποιούνται σιδηροδρόμοι περισσότερο σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ Μάικελ. Κύριος Φακ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχει τονιστεί το θέμα αυτό πάντα. Περισσότερη Ευρώπη ή λιγότερη Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι όλοι μας οι συνάδελφοι υποστηρίζουν την περισσότερη Ευρώπη και γι' αυτό εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο Μπράιαν Σίμψον ότι χρειαζόμαστε την πλήρη διαλειτουργικότητα να ξεπεράσουμε όλα τα τεχνικά εμπόδια και φραγμούς, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα να μιλάμε για ανταγωνισμό. Γι' αυτό και εγώ συμφωνώ για το ότι αυτές οι τρεις προτάσεις, και μιλάω τώρα για τις τρεις εκθέσεις, Πιλμπά, Μπαραντίκα, ε, Κράμερ και Τσίλε, Ζήλε, να αντιμετωπιστούν από κοινού γιατί είναι μεγάλη σημασία για την πρόοδο στο συνδρομικό τομέα. Συγκεκριμένα για την έκθεση του Μίκαελ Κράμερ. ε, όπως τόνισε χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο ασφάλειας ή σιδηρόδρομοι και θέλουμε να το διασφαλίσουμε και για το μέλλον και αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει και κατά τη διάρκεια της του σιδηροδρομικού τομέα. Εξακολουθούμε βέβαια να έχουμε πάρα πολλούς φορείς οι οποίοι εμπλέκονται. Υπάρχει χρήση και καταφυγή πολλών υπεργολάβων που δεν έχουν όλη την δυνατότητα να εξασφαλίσουν το ίδιο επίπεδο ασφάλεια και συγχρόνως αυξάνεται και η σιδηροδρομική κίνηση, κάτι το οποίο δεν είναι αρνητικό αλλά θετικό. Γιατί η κυρία, η κυρία Μπιρμπάου έθεσε ένα παράδειγμα για, τις, ε, για την κίνηση από το Βέλγιο στο Λουξεμβούργο, όπου το Λουξεμβούργο δεν αποδέχεται την πιστοποίηση των φρένων στο Βέλιο. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι η πολυπληθώρα των εμπλεκομένων και πώς μπορείς κάτι το οποίο έχει λειτουργήσει σε επίπεδο ικανοποιητικό για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να τροχοπεδηθεί από έναν άλλο φορέα. Γι' αυτό εγώ θέλω να χαιρετήσω και τις προτάσεις των διαφόρων εισηγητών να συνεργαστούν από κοινού οι τρεις εκθέσεις να προχωρήσουν παραλλήλως, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και πάλι στην έκθεση Κράμερ. Η μείωση του αριθμού των εθνικών κανόνων είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια, αλλά και μεγαλύτερη συνεκτικότητα των κανόνων μεταξύ τους. Και επίσης θα πρέπει να είναι σαφής ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών. Εκεί η Κομισιόν πρέπει να είναι πιο σαφή στην πρότασή της. Να υπάρχει λοιπόν η συνεργασία μεταξύ των εθνικών και των ευρωπαϊκών φορέων, αλλά να υπάρξει σαφής οριοθέτηση των ευθυνών ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη. Το εθνικό επίπεδο ασφάλειας θα πρέπει να παραμείνει, δεν θα πρέπει να ενοποιηθεί προς τα κάτω και επίσης οι κανόνες οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε σχέση με την συντήρηση του τροχαίου υλικού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δεν έχω μεγάλη σαφήνεια για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά θέματα, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ στενά συνδεδεμένα με την εξασφάλιση της ασφάλειας. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο, ο σωστός έλεγχος του χρόνου ε, εργασίας και του χρόνου ανάπαυσης είναι απαραίτητος και στον τομέα αυτό και μια λεπτομέρεια που είναι σημαντική όμως αφορά το άρθρο 10 η δυνατότητα να υπάρχουν κοινά πιστοποιητικά ασφάλειας και εδώ θα πρέπει να έχουμε και μια μεταβατική περίοδο και επίσης αυτό που αναφέρθηκε η δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας για παραβίαση κανόνων. Υπενθυμίζω αυτά τα οποία είπε η Κριστίντα Ιβεράκ χθε για τις αεροπορικές μεταφορές. Ήταν πράγματι και εκεί πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Αϊάλα για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, ακόμα και αν έχουμε κάποιες διαφορές. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό να ενισχύσουμε το ρόλο και την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, να ενισχυθεί το θέμα της ε, άδεια ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, ο κίνδυνος ποιος είναι. Είναι αν δεν είναι ξεκάθαρο το επίπεδο ευθυνών του καθενός. Τι κάνουν οι εθνικές υπηρεσίες, για παράδειγμα, οι εθνικές ε, αρμόδιες αρχές. Γιατί ακούμε διάφορα ε, για το πακέτο αυτό, ότι υπάρχει ο πειρασμός από τη στιγμή που δίνει τις άδειες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, οι εθνικές αρχές να μην έχουν πια καμία ευθύνη. Μίκαελ, θα πρέπει να διασφαλίσουμε το επίπεδο ευθύνη του καθενό. Παρόλο που ενισχύουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων και του επιτρέπουμε την πιστοποίηση κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εθνικές αρχές δεν έχουν καμία ευθύνη. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Γιατί μπορεί να υπάρξει και θέμα επικάλυψης, αλλά μπορεί να υπάρξει και το αντίθετο. Δηλαδή, ο καθένας να θεωρεί ότι δεν είναι δικιά του η αρμοδιότητα. Και έτσι όταν προκύψει πρόβλημα, αντί να δούμε ποιος ευθύνεται. Όσον αφορά τώρα τις υποδομές. Αντιλαμβάνομαι και εγώ ότι υπάρχει τάση οι εθνικές αρχές να κρατήσουν την αρμοδιότητα για την απόφαση, αλλά μερικές φορές λέμε ότι τα θέματα καλά δεν τα ξέρουν οι εθνικές αρχές, τα ξέρει μόνο ο ντόπιο, ε, τέσσερα χιλιόμετρα από το χωριό, παραπέρα δεν ξέρει κανείς τίποτα. Δεν είναι δυνατόν όμως να έχουμε 28 διαφορετικά ε, συστήματα επειδή οι αρχές στην κάθε περιφέρεια θα αποφασίζουν για τα δικά τους μέτρα και σταθμά. Άρα επικουρικότητα, προσοχή. Με τόσα λεφτά μάλιστα που πηγαίνουν από ευρωπαϊκά κονδύλια πρέπει ακόμα και αν υπάρχουν πολλές αρχές ένας να έχει την ε, τελική αρμοδιότητα και την ευθύνη. Για την τροπολογία 24 τώρα, Μίκαελ, λες κάτι που εμφανίζεται και στην έκθεση για τη διαλειτουργικότητα είναι κάτι που υπάρχει στην Γερμανία, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω πολύ καλά. Ότι υπάρχουν κάποια τρένα δηλαδή που είναι διαπεριφερειακά, κάποια λόγια. Εγώ δεν καταλαβαίνω ακριβώ τι θέλει να πει με αυτό για τη μείωση τη ασφάλεια. Και τι θα κάνουμε με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Γιατί και εδώ υπάρχει κάποια σύγχυση για το πώ θα ελέγχουμε τι θα γίνεται μετά από τη στιγμή που υπάρχει μια κατεξουσιοδότηση πράξη. Ευχαριστώ. Πανιόν, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ. Μάικλ, ευχαριστώ. Το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσής σου με βρίσκει σύμφωνο. Έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά εντοπίζοντας τις ευθύνες, τις αρμοδιότητες, πολύ καλή δουλειά. Ώστε οι καθυστερήσεις να είναι όσο γίνεται πιο λίγες και πιο μικρές. για τον ρόλο των εθνικών αρχών, πως αυτός μειώνεται σιγά σιγά κλπ. Ωραία αυτά. για το πιστοποιητικό ενιαίας ασφάλειας, το ενιαίο δηλαδή πιστοποιητικό αυτό. Αν αρχίσουμε να έχουμε ένα σύστημα ιδιαίτερα περίπλοκο, δεν θα πετύχουμε την ενιαία αγορά που όλοι θέλουμε. Υπάρχουν κάποιοι τομείς αβεβαιότητας κατά τη γνώμη μου. Τι εννοούμε με το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ε, που επεκτείνεται γεωγραφικά. Το ορίζουμε. Αν έχουμε διαφορετικές υποδομές μέσα στην ίδια περιοχή. Μπορεί να υπάρχει ένα συμβατό δίκτυο ή υψηλής ταχύτητας. Έχει σημασία δηλαδή όχι μόνο ο γεωγραφικός χώρος αλλά και η υποδομή. Για τις άδειε όσον αφορά τις υποδομές προτείνονται οι εθνικές αρχές αλλά όταν έχουμε διασυνοριακές υποδομές και στην Ευρώπη συμβαίνει συχνά και θα συμβαίνει ακόμα περισσότερο στο μέλλον κυρίως με τις γραμμές υψηλής ταχύτητας οι διασυνοριακές αυτές υποδομές να θεωρούνται μια ενιαία μονάδα και να μην διαχωρίζονται στα σύνορα. Ιδίω όταν πηγαίνουν υψηλέ ταχύτητε στα τρένα δεν μπορεί να υπάρχει κάτι διαφορετικό στα σύνορα, να αλλάζει. Για τις σχέσεις τώρα των ερευνητικών αρχών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού υπάρχουν περιπτώσεις που να μην γνωρίζει την κατάσταση ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός και να πρέπει να βοηθήσουν οι εθνικές αρχές. Μην υπάρχει εδώ σύγκρουση συμφερόντων. Η ιδέα της κυρίας Μπιλμπάου τώρα για έναν κώδικα καταχώρησης των στερεοδρομικών οχημάτων μου άρεσε. είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε την ασφάλεια από τον κοινωνικό ρόλο, τους κανόνες αυτούς. Αν βέβαια αρχίσουμε να είμαστε περιγραφικοί, θα καταλήξουμε σε ανόητα πράγματα. Γιατί αν έχει ένα νυχτερινό τρένο δηλαδή και ξεπεράσει τα 10 λεπτά, τι θα πεις. Α, εδώ σταματάμε και δεν θα προχωρήσει τα επόμενα 10 λεπτά. Πρέπει να υπάρχει κάποια ευελιξία δηλαδή στο καθορισμό των ορών εργασίας, ορών οδήγησης. Αλλιώς θα μπλοκάρει το σύστημα παντελώς. Κύριε Ζήλε, τέσσερα λεπτά κι εσείς. Ευχαριστώ. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και εγώ τον Μίκαλ για... Να τον ευχαριστώ για την πρότασή του Τώρα μερικά στοιχεία που θα, στα οποία θα ήθελα να αναφέρω τώρα για το ενίο πιστοποιητικό ασφάλειας ε, θα πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η πρότασή του σε κάποια στιγμή θα καταργηθεί και θα χρειαστούν περισσότερες απαιτήσει και πιστεύω πως ε, αυτό το πρώτο τμήμα θα συνεχίσει να ισχύει ακόμα και αν το ενίο πιστοποιητικό χρειαστεί να εγκριθεί από τον, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Φυσικά οι σιδηροδρομικές εταιρείε δεν θέλουν να λειτουργούν σε ένα μόνο κράτος. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το κόστος που χρειάζεται για αυτήν την προσαρμογή. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι όταν μιλούμε για ενδιαφερόμενους θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το ενδιαφέρον, το συμφέρον αυτών των ε, οργανώσεων, των επιχειρήσεων. Συμφωνώ με τις προθεσμίες ε, των τριών μηνών μετά από την υποβολή της αίτησης, αλλά με απασχολεί το ζήτημα των ε, ενός ή δύο ετών μόνο εάν είναι διατεθειμένες οι εταιρείε να το πετύχουν μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να ισχύσει, αλλά αυτό θα πρέπει να εξεταστεί. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να γνωρίζουμε ποιος είναι αρμόδιος για τη λήψη των αποφάσεων. και να μην οδηγηθούμε σε συγκρούσεις συμφερόντων. Και τέλος, να πω ότι με ανησυχεί το σύστημα όπου ανωνύμως μπορεί κανείς να κοινοποιεί ενδεχόμενες ε, απειλές για ζητήματα ασφάλειας. Εάν ε, δεν είναι ανώνυμες τέτοιους καταγγελίες, ε, τότε θα μπορέσουμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Τώρα, Το ε, ανώνυμες κοινοποίησεις ε, νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος τρόπος ε, για να βελτιώσουμε την ασφάλεια. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόβατσεκ, τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα τα χρειαστώ αυτά τα τέσσερα λεπτά. Να υπογραμμίσω ότι Όλοι οι συναδελφοί μου απατώνται ολίγων αν θεωρούν ότι υπάρχει μονάχα ένας φορέας πιστοποίησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει ότι αυτός ο ένας φορέας θα μπορέσει να εξασφαλίσει και τους κανόνες ασφαλείας και ότι με τον τρόπο αυτό θα λύσουμε το πρόβλημα. Φοβάμαι ότι ο φορέας αυτός θα είναι τρομερά απασχολημένος, θα χρειαστεί περισσότερο προσωπικό, περισσότερο χώρο, χρηματοδότηση και αυξημένο προϋπολογισμό. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για την διαλειτουργικότητα. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια ενιαία νομοθεσία και ένα ενιαίο σύνολο κανόνων. Υπάρχουν διαφορετικές ηλεκτρικές μηχανές έλξης και υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές ε, προδιαγραφές σε ό,τι αφορά το τροχαίο υλικό. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων ασφαλείας και μόνο να υπάρχει ένα σώμα το οποίο θα ερμηνεύει αυτούς τους κανόνες. Και με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να καλύψουμε όλες τις μηχανές και το τροχαίο υλικό. Αλλά δεν μπορεί αυτό να γίνει το έργο μόνο από ένα φορέα. Δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αυτόν τον τεράστιο φόρτο εργασίες. Επομένως, για μένα από τη μία πλευρά θα πρέπει να υπάρχει το ενιαίο αυτό πλαίσιο κανόνων που είναι απαραίτητο για να υπάρξει ενότητα στο ευρωπαϊκό συνδυοδομικό σύστημα, ενιαίοι κανόνες ασφάλειας, ενιαία διαδικασία πιστοποίησης κτλ. Αλλά παράλληλα θα πρέπει να διευκρινίσουμε ποιος θα ελέγχει την εφαρμογή αυτών των κανόνων και ποιος θα τους εφαρμόζει. Εδώ ο Ευρωπαϊκός Φορέας Σιδηροδρόμων θα πρέπει να αναλάβει την εποπτεία της εφαρμογής των κανόνων αυτών και την εξασφάλιση του σεβασμού τους. Τότε όλα αυτά τα πιστοποιητικά μπορούν να είναι διεθνούς χαρακτήρα, πανευρωπαϊκού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για υποδομές, είτε πρόκειται για τροχαίο υλικό. Αλλά αυτή τη στιγμή μόνο οι δισελομηχανές μπορούν να διασχίζουν όλη την Ευρώπη. Έχουμε μονάχα τρεις τύπους μηχανών που είναι γενικά πιστοποιημένες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανένας να διασχίσει όλη την Ευρώπη με μία μονάχα μηχανή. Και επίσης η έρευνα των ατυχημάτων για τα ατυχήματα πρέπει να γίνεται με ένα υπεύθυνο τρόπο και να είναι και έγκαιρη η έρευνα αυτή. Επίση, επίσης όλες οι διαβάσεις μεταξύ δρόμων και δρομικών γραμμών είναι οι χώροι όπου γίνονται πολλά ατυχήματα και συνήθως αυτά τα ατυχήματα οφείλονται στο γεγονός ότι τα αυτοκίνητα δεν σέβονται τους κανόνες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζασάδα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θέλω να απαντήσω λίγο στο θέμα της αποκλειστικότητας του ενιαίου δηλαδή πιστοποιητικού που θα εκδίδει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Επί της αρχής νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα. Αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε κάποιες ιδιαιτερότητες που ίσως να πρέπει να οδηγήσουν σε εξαιρέσεις. Σε ορισμένες χώρες μέλη, για παράδειγμα, όπου υπάρχουν εξωτερικά σύνορα με τρίτες χώρες, συνδέονται με διαφορετικό τρόπο με αυτές και αν θα θέλαμε να ακολουθήσουμε αυστηρά τους κανόνες, τότε οι τροχές της τρίτης χώρας κανονικά δεν θα έπρεπε να μπορούν να μπουν στην λόγο ευρωπαϊκή χώρα. Νομίζω λοιπόν ότι οι εθνικές αρχές των λόγω χωρών μελών θα πρέπει να μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά για τέτοιου είδους ε, υλικό τροχιάς. Θα μπορούσα εδώ να απαντήσω και σε άλλα σχόλια του κύριου Ζήλε για παράδειγμα ότι η εποπτεία είναι μια καλή ιδέα και ο έλεγχος, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρχει περιθώριο για εξαιρέσεις, αποκλήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη διαλειτουργικότητα. Ίσως και εκεί να υπάρχει περιθώριο για εξαιρέσεις επειδή υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε πολλές χώρες μέλη. Και ένα σχόλιο ακόμα. Για τη μεταβατική περίοδο. Ίσως να μην είναι αρκετά μεγάλη, ίσως θα έπρεπε να είναι πιο μεγάλη μεταβατική περίοδος για να προλάβουμε να προετοιμαστούμε και καλύτερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πακέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πάλι ευχαριστώ τον εισηγητή για τη τόσο φιλόδοξη έκθεσή του η οποία ξεπερνά και την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη βελτιώνει θα έλεγα. Γι' αυτό ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Η παρουσίαση που κάνατε βάζει την ασφάλεια στα σωστά πλαίσια, ότι δηλαδή καμία παραχώρηση για θέματα ασφάλειας. Από την άλλη μεριά οι συνδρόδρομοι πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικά. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ που το παρουσιάσατε έτσι. Ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης, όπως και με τη διαλειτουργικότητα, έτσι και τώρα, ήταν το θέμα της διάρθρωσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού με τις Εθνικές Αρχές. Ε, προτείνατε, μάλιστα, Πρόεδρε, κάποια διάρθρωση ανάμεσα και στις τρεις εκθέσεις. Σωστό. Για την ασφάλεια Πάντως υπάρχει ένα σημείο το οποίο θα μπορούσαμε να υπογραμμίσουμε και αυτό είναι ότι αν όπως προτείνεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός εκδίδει τα πιστοποιητικά, τότε οι εθνικές αρχές θα μπορούν να ελέγχουν τα διάφορα τμήματα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα βελτιωθεί η διαχείριση του συστήματος, κάτι το οποίο είναι θετικό ως εξέλιξη. Και κάποια τώρα ειδικότερα σχόλια για τις τροπολογίες που μιλούν για την διαφάνεια και για αυστηρές προθεσμίες. Συμφωνώ, είναι μια συζήτηση που κάναμε και πρόσφατα, ναι, πολύ χρήσιμο. Για τη μεταβατική περίοδο να περιοριστεί στον ένα χρόνο, έχω το ίδιο σχόλιο όπως έκανα και πριν για την έκθεση της κυρίας Μπιλβάου. Δηλαδή, από μπορεί να είναι λειτουργικό, αλλά όσον αφορά την ε, διοργανική διαδικασία, δεν ξέρω. Τώρα για τους ορισμούς, ίσως θα έπρεπε να φροντίσουμε να είναι όπως και στην έκθεση για τη διαλειτουργικότητα. Να μην υπάρχουν αποκλήσεις. Κάτι ακόμα, ο εισηγητής προτείνει ένα σύστημα επικοινωνίας ώστε να αναφέρονται περιπτώσεις που ίσως οδηγούν σε κίνδυνο με διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο και να υπάρχει μια κεντρική τράπεζα δεδομένων όσον αφορά τα ατυχήματα και τα διάφορα συμβάντα, όπως συμβαίνει και με την αεροπορία. Ναι, αλλά πρέπει να δούμε τους πόρους τότε κάτι το οποίο θα αξιολογηθεί στο τέλος της διαδικασίας για να δούμε αν μπορούν να βρεθούν οι κατάλληλοι πόροι. Είναι θέμα δημοσιονομικών προτεραιοτήτων. Ένα σχόλιο επίσης για τον ερευνητικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Εδώ όντως υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για κάποιον ο οποίος διαχειρίζεται ένα σύστημα και ερευνά και την ασφάλεια. Το ερευνητικό σώμα, όπως συμβαίνει με την νομοθεσία μέχρι τώρα παραμένει εθνική αρμοδιότητα και το επιβλέπει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός. Θα μπορούσαμε όμως να το συζητήσουμε παρετέρω, άμα θέλετε, με τους σκιώδες και τον εισηγητή. Ο κύριος Μπενιόν αναφέρθηκε και στις διασυνοριακές υποδομές. Ναι, συμφωνώ. Και το ότι θα υπάρχουν όλο και περισσότερες διασυνοριακές υποδομές είναι αλήθεια. Το βλέπετε κι εσείς το έργο σας όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα και για τους χρόνους οδήγησης, ναι, ξέρω ότι είναι σημαντικότερη τροποποίηση αντί για να έχουμε νέους κανόνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Επόμενο θέμα. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Α, όχι. Ναι, σωστά. Μίκαελ, πρώτα να απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Βλέπω ότι έχουμε πολλά κοινά στοιχεία. Αλλά δεν λέω ότι θέλουμε ένα ευρωπαϊκό φορέα που να αποφασίζει για όλα. Όχι, πρέπει να κρατήσουμε τις αρμοδιότητες τους οι ευρωπαϊκοί φορείς. Δεν πρόκειται να κάνουμε ένα τεράστιο τερατώδιο οργανισμό που θα τα καλύψει όλα. Γι' αυτό είναι απαραίτητο η συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορέων να παίξει τον αποφασιστικό ρόλο. Αλλά κάποιος θα πρέπει να έχει τον αποφασιστικό ρόλο για να υπάρχει μια ευρωπαϊκή δομή και να μπορούν οι βιομήχανοι να κατασκευάσουν από τη βάση ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Περί, του τούτου πρόκειται. Ο Ρόμπερτ αναφέρθηκε στις εξαιρέσεις και αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό το οποίο λέει η κυρία Γιάλα Σέντερ. Στην Κάτσρουε υπάρχει, στην Κατσού υπάρχει ένα ε, τραμ το οποίο λειτουργεί μαζί πάνω στις γραμμές των τρένων και μπορεί κανείς να περάσει από το τρένο στο τραμ αυτό. Αυτό είναι πολύ καλό. Μεταξύ του Σάρμπρουκ και του Σάρεμπρουκ υπάρχει επίσης μια τέτοια, συν, ε, μια τέτοια γραμμή η οποία λειτουργεί εν μέρη στο κομμάτι του, του γερμανικού σιδηροδρόμου και μετά στο τμήμα των γαλλικών συνδεδρομών. Όλα αυτά είναι εξαιρέσεις, όλα αυτά μπορούμε να τα ρυθμίσουμε, αλλά αυτές είναι γεωγραφικές ή περιφερειακές εξαιρέσεις, αλλά δεν, έχουν, δεν πρέπει να έχουν εθνικό χαρακτήρα. Η Γαλλία έχει δύο διαφορετικά συστήματα, δεν μπορεί καν να παίρνει εθνικές αποφάσεις γιατί υπάρχουν δύο εθνικά συστήματα. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι τα προβλήματα που βρίσκονται. Δεν υπάρχει παραγωγικά δυνατότητα σύνδεση Εστονία-Λετωνία γιατί είναι διαφορετικά τα συστήματα. Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε ότι οι αποφάσεις είναι στο 95% εθνικές αποφάσεις και τα κοινωνικά θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Για. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε οι φορείς, η Ευρωπαϊκή, να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός φορέας να πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις. Φυσικά μπορεί να έχει συμφωνίες με τους εθνικούς φορείς ασφάλειας, αλλά χρειαζόμαστε να έχουμε και τη δυνατότητα αυτή. Για τα συμβάντα και τα ατυχήματα. Ξέρουμε ότι για πολλά από αυτά τα ατυχήματα υπάρχουν οι εθνικές αρχές οι οποίες προσπαθούν να μην δημιουργήσουν ζημία στους ε, σιδηροδρόμους, στους εθνικούς και κουκουλώνουν πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει όμως να υπάρξει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα ελέγχει που υπήρχαν τα προβλήματα, που υπήρξαν τα ασφάλματα και πρέπει να έχει τις απαραίτητες αρμοδιότητες αυτή η αρχή. Όχι να κουκουλώνεται τα πράγματα. η βάση για να μην επαναληφθεί ένα ατύχημα είναι να υπάρχει η σωστή ανάλυση των αιτιών του. Δεν πρέπει να λέμε ότι Α, αυτό είναι εθνικό ατύχημα, επομένω θα το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Με τον τρόπο αυτό δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά. Γι' αυτό η ΕΡΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ιδροδόμων, θα πρέπει να είναι η γενική, η βασική αρχή η οποία θα εξασφαλίσει τον έλεγχο σε περιπτώσεις ατυχημάτων. Και πολλές φορές υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν την επαρκή εμπειρία και μπορεί αυτή να γίνεται από κοινού από ένα ε, κεντρικό φορέα. Ο Ρόμπερ τώρα για τον κεντρικό φορέα. Θέλω να πω καταρχήν ότι προφανές είναι ότι πολλές από τις τροπολογίες μου πρέπει να ενσωματωθούν, να συγκεντρωθούν μαζί. Σχετικά με τις αρμοδιότητες, όταν ε, ξεκίνησα την εξέταση, θέλησα να αφήσω τον οργανισμό εκτός. Αλλά το ζήτημα είναι, ε, μπορεί να υπάρξει αποκλειστικότητα, γι' αυτό λοιπόν η προσέγγιση μου δεν είναι αποκλειστική, αλλά αφορά διάφορα στάδια. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα των υποδομών. Φυσικά θα πρέπει να χορηγούν οι κατάλληλες Τώρα το θέμα της ασφάλειας και τα σχετικά πιστοποιητικά, όπως ήδη προείπα, θα πρέπει τα πιστοποιητικά αυτά να μπορούν να ισχύουν για το, σε επίπεδο ευρωπαϊκού οργανισμού τώρα για το τροχαίο υλικό και για τις ε, ε, μηχανές έλξης ε, θα πρέπει να υπάρχουν ειδικέ ειδικά βιστοποιητικά. Αυτό είναι απαραίτητο, αλλά χρειάζεται να είναι ενιαία. Στην Ανατολική Ευρώπη είναι πολύ καλά σε κάποιες περιπτώσεις ενσωματωμένα και οι οργανισμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί. Ένα άλλο πρόβλημα που είδα είναι πως ε, στον προτινόμενο κανονισμό δεν ε, αναφέρεται το ζήτημα της ε, χρηματοδότησης ε, και της και του κατάλληλου προσωπικού, δηλαδή της τελέχωσης της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συντηροδρόμων. Απόψή μου είναι οι ενδιαφερόμενοι να αντίχουν τις δυνατότητες των καλύτερων ευκαιριών. Γι' αυτό λοιπόν η ΕΡΑ, ο Εθνικός Οργανισμός, είναι καταλληλότερος από τους εθνικούς οργανισμούς. Αλλά όπως σας είπα επιθυμώ η πρότασή μου να μην αποτελέσει υποβάθμιση της ε, ισχύουσας κατάστασης αλλά βελτίωση. Κάτι ακόμα θα ήθελα να αυξηθεί η ευθύνη της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συντεροδρόμων. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια που καλύπτουν τους εθνικούς οργανισμούς και τον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα της αστικής ευθύνης σε περίπτωση πρόκλησης ε, κάποιων ζημιών. θα πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα φυσικά της αμοιβαιότητας και της πρόβασης της αγορές ε, τρίτων ε, κρατών, ο πλευράς τρίτων κρατών. Στην ε, Ανατολική Ευρώπη και στην ε, στην Βόρειο Ευρώπη, Φιλανδία λοιπά, Η κατάσταση είναι ιδιάζουσα και οι σχετικές ε, πληροφορίες δεν κοινοποιούνται στους άλλους εθνικούς οργανισμούς Φυσικά το ζήτημα είναι ακόμα πιο παράδοξο για τους ε, μηχανές έλξης ε, που δεν μπορούν να περάσουν τα σύνορα. εάν υπήρχε, υπήρχε περίπτωση όπου ο πρόεδρος της Εστονίας θέλει να μεταβεί από την ε, χώρα του στην γειτονική ε, δεν μπορούσε να μεταβεί με τον ίδιο σιδηρόδρομο ενώ θα, θα το αντίθετο εάν ήθελε να μεταβεί στην Ρωσία, στη Μόσχα. Τώρα το ζήτημα της ε, γλώσσας ε, είναι πολύ λεπτό, αλλά αν κάποιος ε, επικοινωνεί σε μια κοινωτική γλώσσα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμο, τώρα θα πρέπει να μπορεί να λάβει την απάντηση στην ίδια γλώσσα. Και δεν νομίζω ότι είναι τόσο δαπανηρό όσο μπορεί κανείς να πιστεύει. Σε κάτω κάτω της γραφής πόσες γλώσσες θα χρησιμοποιούνται. Ευχαριστώ. Ντομινίκ, ε, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Ρομπέρ. Ε, είναι πάντα ευχάριστο να δουλεύει κανείς πάνω σε μια δική του έκθεση. Να κάνω λοιπόν μια μουσική σύγκριση. Το ευρωπαϊκό κοντσέρτο της ε, Ισπανίας, της Ευρώπης ε, νομίζω ότι θυμίζει μια ορχήστρα η οποία αποτελείται από 28 μουσικούς αλλά δεν έχει διευθυντή ορχήστρας. Νομίζω ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να γράψουν ε, τον, την μουσική και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία να την συντονίσει, να παίξει το ρόλο διευθυντή. Υπάρχουν ε, ε, τέσσερις υπηρεσίες. Ε, μία δημιουργεί κάποιες αφιβολίες στο ζήτημα της της καταγραφής και καταχώρησης στο Μητρό δεν είναι κάτι που αμφισβητείται. Τώρα το έλεγχος και η αρρωγή από διάφορους οργανισμούς ε, όπως οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, οι εθνικές αρχές κλπ. Ε, δεν αφισβητούνται εκεί όμως όπου το πράγμα κολλάει είναι η πιστοποίηση διότι εδώ έχουμε κάποιες πράξεις δεσμευτικές και νομίζω ότι ακούσαμε ποικίλε απόψεις. Πιστεύω ότι η αθερίδα θα πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή υπηρεσία. Διαφορετικά δεν έχουμε καμία δυνατότητα να πετύχουμε την ευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα. Αυτό που δεν μπορούμε να αφισβητήσουμε είναι το ενίο ψωπητικό, το ζήτημα του είδου του τροχαίου υλικού. Τώρα για την για τους εθνικούς κανόνες και τους περιφερειακούς κανόνες ε, φυσικά οι εθνικοί οργανισμοί μπορούν να παίξουν ένα διαμεσολογητικό ρόλο αρκεί να ζητήσουν την άδεια της Ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να παρέχουν βοήθεια, αρρωγή, στήριξη Διαφορετικά θα είναι σαν να επαναχωρούμε σε όλα τα ζητήματα της ε, διαλειτουργικότητας ε, και θα έχουμε τους εθνικούς κανόνες, ε, τις προσπάθειες θέσης στην αγορά σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούμε να πιστέψουμε λοιπόν ότι οι λειτουργίες οι εθνικές και οι περιφερειακές θα μπαίνουν περιοριζόμενες τώρα για τις καθυστερήσεις νομίζω ότι είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε, σε όλους ότι μπορούν να έχουν δυνατότητες προσφυγής σε κάποιες ε, διεξόδους, δεν πρέπει να δημιουργήσουν μια κατάσταση αντιμπέριου. Θα ήθελα να επιμείνω λοιπόν στα θέμα του καθεστώτος του προσωπικού και της ΕΜΒΕΣ. Νομίζω ότι το ύψος των χρηματοδότησης δεν είναι ικανοποιητικό. Δεν μπορεί να ζητάμε από την υπηρεσία να ε, κάνει όλα όσα, τις, όσα απαιτούνται, διότι δεν έχει τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για τις αμοιβέ του προσωπικού. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό, διότι ενδέχεται να έχει επιπτώσει στην αποτελεσματικότητα τη λειτουργικότητα, στην διατήρηση και εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και το καθεστώς του προσωπικού αλλά και το ζήτημα της ε, πρόσληψης. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι στο ύψος των δυνατοτήτων των οργανισμών. Θα πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα της περαιτέρω συνεργασίας. Τώρα για το γλωσσικό καθεστώς, εάν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλες οι γλώσσες της Ένωσης, δεν θα το καταφέρουμε και να καταλήξω η μεταβατική περίοδος. Ε, κοιτάξτε, ακούω ανθρώπους που λένε ότι θα πρέπει να περιοριστεί, θα πρέπει να, άλλοι λένε να πρέπει να επιμηκυνθεί. Όλα αυτά συνδέονται με τα μέσα που θα αποκτήσει η Ένωση. Αν έχουμε πολλά μέσα, τότε η περίοδος ε, μεταβατική θα πρέπει να είναι σύντομη θα, και μπορεί να είναι σύντομη. Εάν είναι περιορισμένα αυτά τα μέσα, τότε η περίοδος αυτή θα είναι πολύ πιο μακρά. Ευχαριστώ κύριο Πανιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως υπεγράμισε και ο Ρόμπερτ στην έκθεσή του, αυτό το ενιαίο σύστημα το οποίο περιμένει από εμά ο συνδρομικός τομέας είναι απόλυτα ε, αναγκαίο και υπενθυμίζω αυτό που παρουσίασε ως ε, ορχήστρα με πολλές παρτιτούρες και χωρίς διευθυντή ο συνάδελφος μας ο κύριος Ρίκε Ακολουθώντας τώρα αυτά που είπε ο συγητής μας, ο Ρομπέρτ Ζήλε, εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι ζητούν μια πιστοποίηση ασφάλειας θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στον Ευρωπαϊκό Φορέα ή στον Εθνικό Φορέα. Αν έχουμε μια μηχανή έλξης που κυκλοφορεί μονάχα στο εθνικό έδαφος αλλά αυτό θα πρέπει να είναι η μόνη περίπτωση όπου θα μπορεί να έχει την επιλογή ο ετούμενος κάποιας πιστοποίησης να απευθυνθεί στον εθνικό φορέα και όχι στον ευρωπαϊκό. Πιστεύω επίσης ότι ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να δώσει πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια σε σχέση με την ποινική ευθύνη του Ευρωπαϊκού Συνδρομικού Φορέα και του προσωπικού του το άρθρο 64 που δίνει ποινική ασυλία στον φορέα αυτό, νομίζω ότι θα δημιουργήσει προσκόμματα στη σωστή ε, διερευνήση ποινικών ευθυνών σε περίπτωση ατυχήματος. Επίσης το γλωσσικό καθεστώς του φορέα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον κανονισμό. Και εδώ συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητή. Αντίθετα λυπάμαι γιατί ο εισηγητής δεν έχει λάβει υπόψη στην εκθεσή του την αναγκαιότητα να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία ο Ευρωπαϊκός ιδροδομικός Φορέας θα πρέπει να ενισχύσει τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες του και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη και η απαραίτητη χρηματοδότηση σε αυτό το φορέα και επομένως να γίνουν όλα αυτά που έλεγε ο συναδελφός μας για την επίτευξη μιας ομαλής μετάβασης. Όλες αυτές λοιπόν οι λεπτομέρειες θα πρέπει να ρυθμιστούν και θα προσπαθήσω να το κάνω με τις τροπολογίες μας. Αυτή τη στιγμή έχει μονάχα κανονιστικό, κανονιστική αρμοδιότητα ο Ευρωπαϊκός Φορέας Σιδηροδρόμων θα πρέπει να αποκομίσει την αρμοδιότητα λήψης απόφασης στον σιδηροδρομικό τομέα και θα πρέπει βαθμία να δημιουργηθεί η απαραίτητη ικανότητα στον φορέα αυτό για να μπορέσει να υπομπιστεί τις νέες αυτός αρμοδιότητες. Αυτός ο μεταβατικός μηχανισμός μπορεί να ακολουθήσει το καλούπι αυτών που έχουν γίνει για τον Ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκό Φορέα Ενέργειας ασφάλεια με κάποιες τροποποιήσεις. Και συμμερίζομαι αυτά που είπε ο Ντομινίκ Ρικέ, ότι χρειάζεται μια καλύτερη διευκρίνηση των αρμοδιοτήτων αυτού του φορέα της χρηματοδότησής της των υλικών και ανθρωπίνων πόρων και των ευθυνών του. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε. Κύριος Μπένιον, τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την, ε, την ορμή που έχουμε δημιουργήσει προς την κατεύθυνση της ενιαίας αγοράς στον σιδηροδρομικό τομέα. Αν επιτρέψουμε τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να παραμείνουν στο εθνικό τους κουκούλι, τότε θα είναι πολύ λίγες επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορέσουν οι οποίες θα ζητήσουν ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το άνοιγμα της αγοράς. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι απόλυτα προτιμότερο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων να είναι ο μοναδικός φορέας ο οποίος δίνει τα ενία πιστοποιητικά του του λεχθέντος όμως. Κατανοώ και συμφωνώ ότι ο Ρόμπερτ έχει παρουσιάσει ορισμένα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση και σε ό,τι αφορά την ευκολία πιστοποίησης για αυτούς τους φορείς που είναι και εξακολουθούν να θέλουν να παραμείνουν κυρίως εθνικού χαρακτήρα. Σε ό,τι αφορά το τροχαίο υλικό, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ευρωπαϊκή διαδικασία πιστοποίηση και όχι μοναχά εθνικές διαδικασίες, γιατί ένα από τα κύρια πράγματα τα οποία θέλουμε είναι να υπάρξει μια ενιαία αγορά για τροχαίο υλικό, να μπορεί να χρησιμοποιείται και δεύτερου και μεταχειρισμένο τροχαίο υλικό το οποίο εξακολουθεί να έχει την αξία του. Για να επανέλθω σε αυτά που είπε ο Ρόμπετ, αυτό το οποίο δεν θέλουμε να κάνουμε, να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο το οποίο απλώς επεκτείνει τα εθνικά μονοπόλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε δυνατότητες επιλογής σε ό,τι αφορά τις διαδρομές για να έχουμε αυτά τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά. Και είναι απαραίτητο να υπάρχει και μια διαφοροποίηση στην τιμολόγηση επί τη βάση της περιοχής χρήσης του υλικού. Αυτό που δεν θέλουμε είναι ο φορέας ο ευρωπαϊκός να καταλήξει σε ένα σύστημα τιμολόγησης το οποίο να βολεύει την SNCF ή την Deutsche Bahn αλλά για μια μικρή εταιρεία η οποία θέλει να λειτουργήσει μονάχα μια γραμμή περιφερειακή για λίγα χιλιόμετρα να μην είναι η κατάλληλη τιμολόγηση. Έχουμε και το πρόβλημα αυτό των διαφορετικών συστημάτων που λειτουργούν στις χώρες της Βαλτικής και έχουμε και το πρόβλημα των πολύ μικρών <clears throat> εταιριών. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε ενιαίο τίμημα για τα πιστοποιητικά. Και η γλώσσα μπορεί να είναι ένα πρόβλημα και πάλι για πολύ μικρές συνδροδομικές εταιρείε. Αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δούμε τη σχέση μεταξύ των Εθνικών Φορέων Ασφαλείας και του Ευρωπαϊκού Φορέα Σιδηροδρομών, ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτές τις εθνικές αρχές ως υπεργολάβου σε ό,τι αφορά την χορήγηση αυτών των πιστοποιητικών. Έτσι λοιπόν μπορούν αυτοί οι εθνικοί φορείς να είναι το σημείο επαφής για τις τοπικές επιχειρήσεις που δεν θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο και να ζητήσουν ευρωπαϊκά πιστοποιητικά. Αλλά τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε μια ευρωπαϊκή διάσταση ώστε οι εταιρείε αυτές που μπορούν και θέλουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες σε άλλες χώρες να μπορούν να λειτουργήσουν και αλλού. Τα θέματα αυτά λοιπόν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, δεν μπορούμε να πούμε απλώς αφήστε τα όλα στον Ευρωπαϊκό Συνδρομικό Φορέα, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων, γιατί μπορεί αυτό να οδηγήσει σε υπερτιμολόγηση, ιδίω για τους μικρούς φορείς. Και επίση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε εμπλέκεται στα θέματα αυτά και θεωρεί ότι ασκούνται διακρίσει εις βάρος του να μπορεί να έχει την δυνατότητα προσφυγή στον Ευρωπαϊκό, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων και φυσικά προσβλέπω στη συνεργασία με τον Ρόμπερτ και τον Μιχάλη και τους άλλους εμπλεκόμενους για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά και νομίζω ότι έχουμε όλη τη θέληση να τα πετύχουμε αυτά. Κράμε τέσσερα λεπτά. Πάλι ο Ευρωπαϊκός Φορέας Σιδηροδρόμων, η ΕΡΑ να είναι ευρωπαϊκός φορέας, να συνεργάζεται όμω με τι εθνικέ αρχέ, όπω είπα και ξαναείπα, 95% των αποφάσεων πρέπει να λαμβάνονται σε επίπεδο εθνικό. Θα πρέπει να λειτουργεί ως επόπτης των εθνικών αρχών. Εγώ συμφωνώ. Ως, όσο παραμένουμε σε επίπεδο εθνικής πιστοποίησης, συνεχίζεται η κατάσταση όπως και τώρα και στο παρελθόν. Και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε καθόλου. Είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτό το λόγο η διευκρίνηση των αρμοδιοτήτων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι. Αν δω τώρα την κατάσταση στις βαλτικές χώρες. Η ίδια, το ίδιο, η ίδια μηχανή μπορεί να κινείται στη Φιλανδία, στη Λετωνία και στη Λουθουανία. Μα είναι κάτι αντίστοιχο με τους ενιαίους εθέρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε ε, διμερείς συμφωνίες όπου υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα. Πετάνε οι Αμερικάνικες εταιρείες στο Παρίσι, πετάνε στο Βερολίνο κτλ. Αλλά εμείς μέσα στην Ευρώπη δεν θέλουμε να υπάρχει κάτι τέτοιο, θέλουμε ο καθένας να κρατήσει την τοπική του αγορά. Και επομένως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πλεονεκτήματα για μια μικρή χώρα σαν τη Λετωνία προκύπτουν μονάχα όταν είναι ένας κόμβος για τις συνδέσεις με τη Ρωσία. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε το στόχο οι βαλτικές χώρες να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ατμομηχανές, τις μηχανές έλξης οι οποίες παράγονται στη Ρωσία να λειτουργούν και στην Ευρώπη. Να μπορεί να φτάσει μια τέτοια μηχανή έλξης και στην ε, Γερμανία. Αλλά ακόμα και αν περιορίζεται αυτό μόνο στην ε, Λετωνία, Εστονία και Λιθουανία και Φιλανδία, αυτό είναι σημαντικό. Να μην λέμε ότι αυτοί, αυτές οι μηχανές δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν πράγματος χάρη στη Φιλανδία. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε να τονίσουμε ότι εδώ έχουμε την Ευρώπη και δεν πρέπει να είναι διμερείς μονάχα συμφωνίες δεν είμαστε οι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά η πιστοποίηση πρέπει να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν οι διαφορές αυτές, όπως έλεγα, με τα τραμ ε, και με άλλες περιπτώσεις που ανέφερα. Δεν θέλω φυσικά να μιλήσω καθόλου για τους ιστορικού χαρακτήρα σιδηροδρόμους. Όλα αυτά πρέπει να τύχουν ειδικών ρυθμίσεων, αλλά καταρχήν πρέπει να είναι όλα ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Νομίζω ότι γενικά έχουμε προχωρήσει τα θέματα αυτά. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τους Σκιώδη και όλους αυτούς οι οποίοι έχουν λάβει μέρο στη συζήτηση και φυσικά ευχαριστώ και την Κομισιόν η οποία μας έχει βοηθήσει στα θέματα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν σα δώσω το λόγο κύριε Κόλτσεκ να υποδεχτούμε εδώ επισκέπτε τη κυρία Κρίσμπεκ από την Ένωση των Ταγκοντάνς από τον Μοζέλα στη Γαλλία. Καλώς ήρθατε εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Ελπίζω να βρείτε ενδιαφέρουσα τη συνεδρίαση. Παρακαλώ κύριε Κόλτσεκ, για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, αλλά θέλω να επανέλθω, επιτρέψτε μου, σε κάποιες τεχνικές πτυχές που νομίζω ότι δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη συνάδελφοι. Αν έχουμε ένα σύστημα. Πώς δουλεύουν οι υποδομές. Έχουμε πολλά τέτοια συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρουμε πόσο διαφορετικά είναι τα αποτελέσματα σε δοκιμές. Αν έχουμε πολλά διαφορετικά συστήματα ηλεκτρικής έλξης, για παράδειγμα, τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά. Οι συνάδελφοι είπαν σωστά ότι αν έχουμε ένα σύστημα ελέγχων και αν εφαρμόσουμε και ένα άλλο, τότε δεν θα καταλήξουμε στα σωστά αποτελέσματα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα ειδικό σύστημα ελέγχου του τροχαίου υλικού και άλλων υποδομών. Δεν είναι πολιτικό το θέμα, είναι εξαιτίας των τεχνικών ε, προδιαγραφών, των τεχνικών στοιχείων που ισχύουν. Πρέπει να έχουμε ενιαίους τεχνικούς κανόνες, λοιπόν. Και αν θέλουμε εθνικές αρχές να προσαρμόζονται και αν θέλουμε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός να ε, το ελέγχει, τότε δεν θα βγούμε ποτέ από το φαύλο κύκλο των εξαιρέσεων και μετά από πολλά χρόνια που έχω περάσει στη βιομηχανία μπορώ να σας πω ότι είναι ανοησία κάτι τέτοιο. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Να πω και εγώ δύο λόγια μετά από αυτά που είπε ο Μάικλ και που βεβαίωσε και ο κύριος Πάκετ ο, για τις εξαιρεσει που θα υπάρχουν στο τέταρτο πακέτο. Εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε και το πρόβλημα που γνωρίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, όπου έχουμε την κύρια γραμμή που κυκλοφορεί και στο ΕΜΕΤΙΕΣ. Και ξέρω ότι η ΦΕΝΤΕΚ με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων συνεδριάζουν για να το λύσουν. Προσπαθώ να δω, υπάρχει επιβεβαίωση για όλα αυτά τα ωραία πράγματα που λέμε ατμομηχανή. Τέλος πάντων. Ο κύριος Πακέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δυνατότητα εξαιρέσεων παραμένει. Την δίνουν τα κράτη-μέλη. Δεν νομίζω ότι με τις εκθέσεις αυτές αλλάζει κάτι. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω πρώτα τον εισηγητή τον κύριο Ζήλη για την έκθεσή του. Εγώ ασχολήθηκα πιο πολύ με τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια, αλλά και η έκθεση του κύριου Ζήλη καλύπτει τα τρία στοιχεία κλειδί, τα οποία είναι η υπευθυνότητα και η αρμοδιότητα, κάτι πολύ βασικό και βέβαια για τις δύο προηγούμενες εκθέσεις. Το δεύτερο θέμα είναι οι προσφυγές. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει καλή διάρθρωση ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και τις Εθνικές Αρχές. Και η ασφάλεια και η δημοσιονομική πόροι. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτά. Τώρα υπάρχουν και κάποια άλλα πιο μικρά τεχνικά ζητήματα πάνω στα οποία θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τον εισηγητή. Τώρα για τη διάρθρωση ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνδρομών και τις Εθνικές Αρχές. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι η νομοθεσία θα πρέπει να θέτει την ευρύτερη αρχιτεκτονική. Από εκεί και πέρα όμως θα έπρεπε και θα υπάρχει μεγάλο περιθώριο για διακανονισμούς ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και τις Εθνικές Αρχές. Το είπε και ο κ. Κράμερ αλλά και άλλοι ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τη δουλειά των Εθνικών Αρχών Ασφάλειας αλλά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων αρμόδιος για την έκδοση πιστοποιητικών, αλλά θα συνεργάζονται με τις εθνικές αρχές. Γι' αυτό και θα πρέπει να μπορεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός να έρχεται σε συνεννόηση με μια εθνική αρχή, με ένα σύνολο, μια ομάδα εθνικών αρχών. Και πράγματι υπάρχουν κάποια περιφερειακά δίκτυα στις βαλτικές χώρες για παράδειγμα που είναι κάπως πιο απομονωμένα και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η διάρθρωση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Θα έλεγα να μην αφήσουμε απ' έξω αυτά τα απομονωμένα δίκτυα από τα ωφέλη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου, όχι αντίθετα να δούμε πώς ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός των θα μπορέσει να δουλέψει μαζί τους και να τους βοηθήσει για αυτή τη ε, σχέση που έχουν με τις γείτονες χώρες τους εκτός Ευρώπης πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα ευχαριστώ να δούμε με τον εισηγητή πώς μπορεί να διατυπωθεί το κείμενο προς αυτή την κατεύθυνση. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ όλους και σας Πρόεδρε για το φιλόδοξο τόνο που πήρε η συζήτησή μας για αυτά τα θέματα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέρφους για τα σχόλιά τους και θα αντιδράσω σε αυτά. Πρώτα απ' όλα για τις μεταβατικές περιόδους. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί πολύ με αυτό. Φαντάζομαι ότι θα έρθουν τροπολογίες και βάσει των τροπολογιών αυτό θα καταλήξουμε σε, ένα καλό συμβιβασμό. Για τις δαπάνες. Πόσο θα ζητά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Αυτό δεν έχει καθοριστεί. Ήθελα να βάλω κάποιο όριο Πάντως, αν βάλουμε αποκλειστικότητα στις υπηρεσίες του Διεθνούς Οργανισμού, αυτό σημαίνει ότι οι σχέσεις με τις εθνικές αρχές δεν ε, διακανονίζονται καθόλου. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η σχέση νομίζω και για τους πολιτικούς θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να εξηγήσει κανείς στους σειροδρόμους του που θέλουν να λειτουργήσουν σε μια εθνική αγορά και επιβατικά τρένα υπάρχουν που λειτουργούν σε μία μόνο χώρα, να πρέπει να πληρώσουν παραπάνω από ό,τι πληρώνουν σήμερα για να έχουν τις ίδιες υπηρεσίες. Ε, πώς θα το εξηγήσετε αυτό στους πελάτες. Θα αυξηθεί η τιμή των εισιτηρίων τότε για τους επιβάτες για να καλυφθεί αυτό το κόστος. Εγώ νομίζω ότι πολιτικά δηλαδή δεν στέκει. Και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να αφήσουμε αυτή την ε, ενιαία θηρίδα για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων μόνο για ό,τι μπορούν να κάνουν καλύτερα και φθηνότερα από ό,τι οι εθνικές αρχές. Αυτή θα πρέπει να είναι η αρχή μας. Για τη σχέση με τη Ρωσία, για παράδειγμα. Πολύ ωραία αν ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων μπορεί με τον κύριο Γιακούνη και τους άλλους να τα βρούνε. Πολύ ωραία. Μακάρι. Ας αφήσουμε λοιπόν την πόρτα ανοιχτή αν η Λετωνία με την Εστονία θέλουν να έχουν μια κοινή επιχείρηση και να έχουν σχέσεις με τη Ρωσία στα πλαίσια των εθνικών τους αρχών, πολύ καλά. Αν πάλι νιώθουν ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ρώμα είναι πιο ισχυρός από ότι ο αντίστοιχος της Ρωσίας, τότε σε έρθουν σε αυτόν. Ας τους αφήσουμε την επιλογή και μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Αλλιώς δεν είναι δυνατόν. Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρομών προσπαθούμε να έχουμε πληροφορίε για το τροχαίο υλικό στη Ρωσία. Ε, δεν μπορούμε, δεν τα καταφέρνουμε. Δεν γίνεται. Αυτά. Πάντω σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλου και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε καλό συμβασμό. Α, ναι, και κάτι τελευταίο. Είπατε, μετά την έκθεση της κυρίας Μπιλμπάου, κάτι για τα, τις τεχνικές προδιαγραφές και διακρίνατε τα τεχνικά στοιχεία από τα πολιτικά. Ε, πολύ σημαντικό. Και εγώ συμφωνώ. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια κενά θέλουμε μεγαλύτερη ελευθέρωση στους σιδηροδρόμους. Αν λοιπόν ο τεχνικός πυλώνας προχωρήσει περισσότερο, ίσως θα πρέπει να προχωρήσουμε και στις άλλες πτυχές. Ευχαριστούμε. Για τις τεχνικές πτυχές, ναι, εντάξει, ξέρω ότι όλοι συνεργαζόσαστε και σκιώδεις, πολύ καλό. Το τελευταίο που θέλουμε είναι να έχουμε μια έκθεση που να λέει ένα πράγμα και μια έκθεση που να λέει κάτι διαφορετικό. Προσοχή λοιπόν. Έτσι, οι τρεις εισηγητές λοιπόν και οι σκιώδεις φροντίστε οι εκθέσεις σας να λένε τα ίδια πράγματα, έτσι. Να υπάρχει μια συνεκτική τελικά τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο τέλος. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών, σας υπενθυμίζω, είναι η 16 Σεπτεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίας. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 26 Νοεμβρίου και στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο του 2014. 16 Σεπτεμβρίου λοιπόν προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 6 η ώρα το απόγευμα. Έτσι εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα το πρωί. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε τον Λιθουανό Υπουργό ε, Μεταφορών, τον Προεδρεύοντα, στις 3. Ας αρχίσουμε στην ώρα μας γιατί θέλουμε μια ώρα για την ανταλλαγή αυτή απόψεων και μετά να περάσουμε στα επόμενα θέματα. Στις 3 λοιπόν.